Και περνάμε στην, στο επόμενο σημείο που είναι η έκθεση της Εύα Μάιντελ επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών. Η κυρία Μάιντελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, φέτος Ερωτάζουμε τα 25 χρόνια από την έναρξη της ενίας αγοράς. Ταυτόχρονα όμως οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη ακόμη δεν μπορούν να αποκομίσουν πλήρως τα ωφέλη λόγω κάποιων φραγμών που συνεχίζουν να υπάρχουν σε διάφορους τομείς. Οι διασυνοριακές πληρωμές είναι σημαντικές για την ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς πολίτες και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών από, τη ζώνη, από τις χώρες εκτός της ζώνης ευρώ συνεχίζουν να έχουν σημαντικές επιβαρύνσεις παρά το ενιαίο ευρωπαϊκό, τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών. Γι' αυτό χαιρετίζουμε αυτή την πρόταση τη Επιτροπής, γιατί θα δίνει τη δυνατότητα στου πολίτες της Ευρώπης ε, να μεταφέρουν χρήματα διασυνοριακά με το ίδιο κόστος όπως θα είχαν για μεταφορά νομισμάτων στο δικό τους νόμισμα. Είναι απαραίτητο να έρθουν οι φραγμοί για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ε, και εκτός της ζώνης ευρώ και αυτό θα βοηθήσει και τον ανταγωνισμό μέσα στη ζώνη του ευρώ. Η Επιτροπή υπολογίζει ότι περίπου 900 εκατομμύρια θα είναι η εξοικονόμηση για τους πολίτες από το μέτρο αυτό. Αποτέλεσμα θα είναι επίσης και πολύ μεγαλύτερη ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευκολότερη ε, κυκλοφορία των υπηρεσιών και των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπάρχει μεγαλύτερη επιλογή των καταναλωτών αφού θα μπορούν να επιλέγουν το νόμισμα στο οποίο θέλουν να κάνουν ε, την ε, μεταφορά. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η εντολή που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για την ανάπτυξη ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων είναι ένα απαραίτητο μέτρο αλλά υπερβαίνει το στόχο του παρόντος κανονισμού. Και η επιβολή ανώτατου του ορίου στο κόστος μετατροπής νομισμάτων ε, θα μπορούσε να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην αγορά. η παρούσα έκθεση αποφεύγει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα γιατί πιστεύουμε ότι δεν ανταποκρίνεται στους στόχους τους οποίους ε, ε, θα θέλαμε. Ε, η εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας είναι εφικτή εφόσον υπάρχουν σαφείς απαιτήσει για τους παρόχους υπηρεσιών. Στόχος είναι να βελτιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής προς την κατεύθυνση αυτή και έχουμε κάνει κάποιες διευκρινιστικές τροπολογίες. Ο κανονισμός αυτός μας δίνει την ευκαιρία να δείξουμε στην πράξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει συγκεκριμένες λύσεις για τους πολίτες της και να αντιμετωπίσει τις ανισότητες στην ενιαία αγορά. Ευχαριστώ ε, και την ομάδα μου και τη γραμματεία για τη δουλειά που έχουν κάνει μέχρι τώρα και έχουμε δεσμευθεί να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους ούτως ώστε να έρθει άλλος ένας φραγμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να έχουμε και καλύτερες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Οι σκιώδεις εισηγητές. Όλοι Λούβιξον για την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Μαϊντέλ, για την έκθεσή της και για τις παρατηρήσεις της. Νομίζω ότι είναι θετικό το ότι και η Επιτροπή και η εισηγήτρια θέλουν να εναρμονίσουν το κόστος για τις διασυνοριακές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα κράτη-μέλη. Ούτως ώστε το κόστος να είναι το ίδιο όπως και για τις ε, μεταφορές μέσα στην ίδια χώρα, στο ίδιο νόμισμα. Αλλά ε, βλέποντας την πρόταση της Επιτροπής, υπάρχουν πολλά τα οποία θα μπορούσαν να συμπληρωθούν. Στο σχέδιο δράσης η Επιτροπή λέγει ότι θέλει να μειώσει το κόστος για τις διασυνοριακές συναλλαγές σε όλα τα κράτη-μέλη. Η εκθέση του Κοινοβουλίου για το σχέδιο δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ζητά από την Επιτροπή να μειώσει και τα τέλη για τις διασυνοριακές συναλλαγές σε όλες τις χώρες. Βάσει των τεσσάρων εναλλακτικών λύσεων της Επιτροπής, οποιαδήποτε αλλαγή του κανονισμού θα σημαίνει ότι θα είναι ίδιο το κόστος για τις διασυνοριακές ε, συναλλαγές όπως και για τις συναλλαγές εντός ενός κράτους μέλους ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο ε, γίνεται η συναλλαγή και ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο γίνεται η συναλλαγή. Αν το κόστος λοιπόν είναι το ίδιο σε όλα τα κράτη-μέλη, ε, οι αλλαγές του κανονισμού θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα νομίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3 δισεκατομμύρια ευρώ νομίζω ότι ε, θα ε, είναι η εξοικονόμηση για τους ε, επενδυτές και τις επιχειρήσεις και 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο η εξοικονόμηση όσον αφορά το όφελος για τους καταναλωτές οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ και οι επιχειρήσει θα πρέπει να υποφεληθούν τα μέγιστα από αυτή την αλλαγή. Σήμερα οι καταναλωτέ πολύ συχνά πρέπει να καταβάλουν υψηλά τέλη όταν κάνουν πληρωμέ σε άλλη χώρα και επιλέγουν να το κάνουν στο δικό τους νόμισμα. Αυτό οφείλεται σε αυτό το οποίο ονομάζεται δυναμική μετατροπή νομίσματος και οι καταναλωτές δεν έχουν σαφή εικόνα του κόστους της συναλλαγής. Η μεγαλύτερη διαφάνεια είναι απαραίτητη και θα πρέπει οι τράπεζε να υποχρεωθούν να ενημερώνουν τους πελάτε για αυτή τη δυναμική μετατροπή νομίσματος, ούτω ώστε οι πολίτες να επιλέξουν με ποιο τρόπο θέλουν να κάνουν τις μετατροπές. Αν θα χρησιμοποιήσουν ε, το δικό του ε, νόμισμα ε, ή αν θα πρέπει η μετατροπή να γίνει μέσω του συστήματος πληρωμών της τράπεζας αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι δυνατόν να τίθενται από τους καταναλωτές ε, όταν ε, θέλουν να κάνουν την ε, συναλλαγή. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και κατά την ανάληψη χρημάτων και κατά την αγορά. Και η τράπεζα που εκδίδει την κάρτα θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη να έχει μεγαλύτερη διαφάνεια και τη στιγμή που γίνεται η συναλλαγή θα πρέπει να μπορεί να ενημερωθεί ο καταναλωτής που θα, κάνει, θα επιλέξει τον τρόπο μετατροπή του νομίσματος, ακόμη και αν καταγραφεί η πληρωμή δύο ή τρει μέρες αργότερα. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο και προσβλέπω στην επικοδομητική συνεργασία με την συγκήτρια την κυρία Μεντέλ για τις επόμενες, κατά τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you for the e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 και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπονται και για τα ανώτατα όρια κόστους της ε, συναλλαγματικής αλλαγής. Είναι λύσεις οι οποίες ε, θα έλεγα εδώ και αρκετό καιρό έχουν ε, υιοθετηθεί Βλέποντας ότι στο παρελθόν υπήρχαν ανώτατα όρια για το κόστος μιας συναλλαγής και αυτό είχε οδηγήσει στην ανάπτυξη της μαύρης, θα έλεγα, της φεάς αγοράς. Τα θυμόμαστε αυτά. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι απαιτείται να υπάρξει μια νέα μορφή συνεργασίας θα πρέπει να μην υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις αδικαιολόγητες όπως το παρελθόν. Το κείμενο στα αγγλικά ε, έχει προκαλέσει κάποια στοιχεία περιέργειας από πλευράς μου. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν το σύνολο των νομισμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βελτιώσουμε τη διαφάνεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα χαιρετήσω και θα υποστηρίξω απόλυτα την πρόταση της Κομισιόν. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα της διαφάνειας στον τομέα των διαμεθοριακών αλλαγών νομισμάτων. Αν αντιμετωπίσουμε συνολικά την ενιαία αγορά, πρέπει να εξασφαλίσουμε ισότητα μεταχείρισης σε όλη την Ένωση. Είναι ευπρόσδεκτη η μείωση του κόστους μεταφορών, χρημάτων, μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ε, βασμάτων σε ευρώ και μη. Και αυτό εξασφαλίζει στους χρήστες πλήρη διαφάνεια όταν πληρώνουν για τέτοιου είδους συναλλαγές. Όσον αφορά το σχέδιο έκθεσης κυρίας Μαϊτέλ, συμφωνώ και εγώ στην θετική προσέγγιση προς το κείμενο της Κομισιόν πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν χρήσιμες προσθήκες όπως η διευκρίνηση που προσθέτει η συγγήτρια με την τροπολογία 10 που εξασφαλίζει ότι θα υπάρξουν εναλλακτικές ε, ε, ε, δυνατότητες στις μετατροπές νομισμάτων προς το χρήστη με τρόπο ξεκάθαρο. Σήμερα έχει κανείς την επιλογή να επιλέξει στο εσωτερικό του νόμισμα που μοιάζει ότι είναι η απλούστερη προσέγγιση. Πιστεύω ότι αν ξεκαθαριστούν το κόστος και οι ισοτιμίες που θα χρησιμοποιηθούν θα ωφεληθούν σημαντικά οι καταναλωτές. Επίσης η συγγήτρια έχει προτείνει να, ε, να αφαιρεθούν το RTS του EBA και να υπάρξει μια μικρότερη μεταβατική περίοδος με τρόπο ώστε να μειωθεί το κόστος προς τις, των επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω και είμαι ανοιχτό για να διερευνηθεί ο καλύτερος τρόπος τόσο για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και προσβλέπω στην μελλοντική συζήτηση των θεμάτων αυτών. Ευχαριστώ. Ε, για την ΚΟΕ λοιπόν ο κύριος Βιέγκας. Nós eh, εμείς είμαστε ευαίσθητοι σε σχέση με τις ανησυχίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί γύρω από την έκθεση αυτή. Όταν κάποιος κάνει μια συναλλαγή με δύο διαφορετικά νομίσματα, πάρα πολλές φορές καλείται να πληρώσει ένα υψηλό κόστος. Ένα άλλο πρόβλημα όμως καθοριστικό για μας είναι το ποσοστό κέρδος των τραπεζών. Στην Ισπανία τα επίπεδα αυτά είναι πάρα πολύ υψηλά και αδικαιολόγητα, ατεκμηρίωτα. Να θυμηθούμε επίσης τις δηλώσεις που είχαν κάνει οι εποπτικές αρχές που έδιναν κίνητρα ουσιαστικά και ευαισθητοποιούσαν τις τράπεζες έτσι ώστε να προσπαθήσουν μέσα από τις χρεώσεις αυτές να καλύψουν τα προβλήματα παραγωγικότητας τα οποία είχαν και κερδοφορίας γενικότερα. Στην Πορτογαλία το κόστος ξεκινάμε από ένα ευρώ ανά συναλλαγή και ανεβαίνουν ε, δυστυχώς ε, πάρα πολύ και φτάνουν και τα 20 ευρώ. Και φυσικά ε, πάνω σε αυτό το κόστος προστίθενται και φορολογίες. Στην ουσία λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει κίνητρα για αυξήσεις του κόστους ενώ μιλάμε για μια <clears throat> θα έλεγα αγορά η οποία λειτουργεί με ολιγοπολιακά κριτήρια. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ανησυχίες και δεν υπάρχουν φυσικά ανώτατα όρια κάτι το οποίο δημιουργεί μια κατάσταση δύσκολη για τους καταναλωτές και μια άλλη ανησυχία η οποία υπάρχει είναι ότι υπάρχουν ορισμένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που εγκαθιστούν μηχανήματα σε διάφορες χώρες και φυσικά κάθε φορά που ε, παίρνει κανείς κάποια χρήματα ε, και έχουν ένα σημαντικό κέρδος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει διαφάνεια σε σχέση με τις επιχειρήσεις αυτές και είναι σαφές ότι ο πολίτης θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για το κόστος. Το θέμα αυτό δεν ισχύει μόνο στην Πορτογαλία. Συνεπώς λοιπόν η πρόταση την οποία έχουμε μπροστά μας είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση αλλά υπάρχουν όπως είπα και αρκετές ανησυχίες που πρέπει να καλύψουμε. Και σύν τις άλλες θα χρειαστούν τρία χρόνια για την εφαρμογή της πρότασης αυτής. Είναι κάτι το υπερβολικό αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να υπάρχει μια τόσο μεγάλη ε, χρονική ε, προθεσμία. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και σε 4-5 χρόνια θα αλλάξει η κατάσταση και δυστυχώς ε, τα συμφέροντα των πολιτών μας θα καταπατηθούν για μια ακόμη φορά. Um, FDD Um...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 κίνδυνος εδώ διασταυρούμενης επιδότησης των τραπεζικών δραστηριοτήτων ε, όταν διαπιστώνουν ότι μπορεί να έχουν κάποιες ζημίες από τις διασυνοριακές συναλλαγές. Ε, και το μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ουσία τεκμηριώνει την επιλογή την οποία έχουν κάνει τα πιστοτικά ιδρύματα και δεν κάνει προτάσεις για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων οι οποίοι δημιουργούνται. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει μια ρήτρα αναθεώρησης ενδιάμεσης και θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή η ρήτρα αυτή να μας δώσει την δυνατότητα στο μέλλον να επανεξετάσουμε τη ρύθμιση έτσι ώστε να ισορροπήσουμε λίγο όλες τις ε, διασυνοριακές συναλλαγές εκεί όπου υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση από το μέσο όρο. Γκίλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Είναι μια καλή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντικό να είναι λειτουργική η εσωτερική αγορά και οι διασυνοριακές πληρωμές ε, να μην κοστίζουν περισσότερο από τις εθνικές. Από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου τώρα φοβάμαι ότι η αποχώρησή μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι οι Βρετανοί πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν τα πλεονεκτήματα αυτών των ε, αλλαγών. Ανησυχώ μάλιστα γιατί οι πρόσφατες δηλώσεις της Βρετανικής κυβέρνησης στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει συμφωνία θα προκαλέσουν ακόμα μερισσότερο κόστος στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και για τη χρήση των πιστοτικών καρτών. Ανησυχώ λοιπόν και για τις εισηγήσεις του τις προτάσεις του εισηγητή μέσω της τροπολογίας υπαριθμών 11. Έχω την αίσθηση ότι σε σχέση με, τις, ε, την μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την Ευρωπαϊκή ε, Αρχή όπως επίσης και οι προτάσεις που γίνονται για την θέσπιση των ορίων έχω την αίσθηση ότι μπορεί και να μην πετύχουν τον στόχο της εύρυθμης λειτουργίας. Απαιτείται διαφάνεια νομίζω έτσι ώστε να, κατανοούν, να κατανοούν οι καταναλωτές το τι ακριβώς συμβαίνει. Κατανοώ αυτούς που λέγουν ότι η αγορά μόνη της μπορεί να κάνει τις απαιτούμενες βροθιώσεις, αλλά μπορεί και να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Θα ήθελα λοιπόν ο εισηγητής ε, να ε, προσπαθήσει να τεκμηριώσει λίγο τις προτάσεις που λέγουν ότι δεν χρειάζεται ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, η Επιτροπή θα ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Χαίρομαι που υπάρχει στήριξη για την πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι θετικό να βλέπει κανείς ότι το πρώτο τμήμα της πρότασης, η εξίσωση δηλαδή του κόστους και των, για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, είναι κάτι το θετικό. Εμείς δεν κάναμε την πρόταση για το σύνολο των χωρών και εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ε, θυμίζω ότι η βασική πρόταση την οποία είχαμε κάνει ήταν πιο φιλόδοξη, αλλά το μέγιστο ποσοστό των συναλλαγών ήδη γίνεται ε, στο ευρώ, με ευρώ ως εκ τούτου δεν υπάρχει δικαιολογία για τα πιστοτικά ιδρύματα να μην χρησιμοποιούν την δυνατότητα αυτή που έχουν για να καλύψουν ένα ίσως μεγαλύτερο κόστος για τις συναλλαγές σε άλλα νομίσματα που είναι μειοψηφικά ουσιαστικά. και νομίζω ότι αν χρησιμοποιήσουν ακόμα περισσότερο το ευρώ και για τις χώρες οι οποίες είναι εκτός ευρώ το κόστος θα είναι ακόμα μικρότερο. Τώρα, ο, ο άλλος στόχος, ε, η διαφάνεια σε περιπτώσεις μετατροπής. Οι τράπεζες προσπαθούν να ανακτήσουν, αν θέλετε, αυτό που θεωρούν απολεσθέν εισόδημα, έσοδο. Ναι με να απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια στην περίπτωση αλλαγής νομίσματος, μετατροπής νομίσματος. Τεχνικά όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητό αυτό. Οι έρευνες που κάναμε δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη να κατανοήσουμε ακριβώς το τι ισχύει σε κάθε χώρα και αυτό θα πρέπει να εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή που είναι σε θέση να το ελέγξει. Η πρόταση που αυτή λοιπόν έχει απορριφθεί από πολλούς και εδώ έχει απορριφθεί επίσης και από την πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου. Εμείς δεν έχουμε εγκαταλείψει την ιδέα, αλλά παρόλα αυτά η πρόταση που γίνεται και από το Συμβούλιο επιτρέπει να σημειωθεί σε ορισμένους τομείς ταχεία πρόοδος όπως επίσης και λήψη περαιτέρω μέτρων, δεν αποκλείεται κάτι τέτοιο, εφόσον αυτά γίνουν δεκτά και από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ε, νομίζω λοιπόν το θέμα είναι να υπάρξουν ωφέλη για τους καταναλωτές, για τους πελάτες των πιστοτικών ιδρυμάτων και νομίζω ότι καλό θα ήταν όπως είπατε και εσείς η διαδικασία να πάει λίγο γρηγορότερα από ό,τι προβλέπετε προς όφελος όλων των εμπλεκομένων. Σας ευχαριστώ η συγγήτρια. Να ευχαριστήσω και εγώ τους σκιώδεις και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο για τις παρατηρήσεις τις οποίες έκαναν και για τη θετική τους ε, με γενικά αντίδραση. Εγώ ε, με πολύ ενδιαφέρον θα συζητήσουμε ε, μαζί, να συζητήσω μαζί σας τις καλές ιδέες που ακούστηκαν εδώ σήμερα. Νομίζω ότι αν και η απόσυρση των εμποδίων στις συναλλαγές ε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πραγματικά ενιαία αγορά για τις ε, λιανικές ε, συναλλαγές. Θα μπορούσε επίσης να ωφελήσει και τις επιχειρήσεις, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην επιβάλλουμε περαιτέρω κόστη διαδικαστικά στις επιχειρήσεις αυτές σε σχέση με συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλό κόστος ορισμένων παρόχων ε, αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες ε, από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί θα αυξήσουν το κόστος άλλων υπηρεσιών για να μπορέσουν να καλύψουν κάποιο πιθανός επιπλέον κόστος. Η πρόταση η οποία προτείνεται εδώ καλύπτει περίπου το 80% των συναλλαγών των διασύνοριακών ε, των ε, ε, κρατών μελών που δεν είναι στη ζώνη ευρώ. Καλύπτουμε λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι σε σχέση με το status quo. Αν δει κανείς το τι έγινε πριν από δύο χρόνια όταν πήραμε την απόφαση για την περιαγωγή ε, βλέπουμε ότι τα επιτεύγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται με πολύ σταδιακό τρόπο και δεν πρέπει συνεπώς να είμαστε ιδιαίτερα ε, βιαστικοί. Η διεύρυνση τώρα της πρότασης αυτή σε όλα τα νομίσματα έχω την αίσθηση ότι είναι ένα απαραίτητο επόμενο βήμα και απαιτείται να υπάρξει πραγματικά μια ουσιαστική ανάλυση των προτάσεων. Όπως επίσης και να υπάρξει και συγκεκριμένη μελέτη των επιπτώσεων που θα προκληθούν από την πρόταση αυτή. Σχετικά τώρα με τις χρεώσεις για τις μετατροπές νομισμάτων, προφανώς και, θα και υπάρχει εδώ ε, χώρος για περισσότερη διαφάνεια. Ελπίζω αυτά τους επόμενους μήνες να γίνουν πραγματικότητα ε, για την λεγόμενη διασταυρώμενη επιδότηση και τις επικαλύψεις ε, εδώ υπάρχει κάποιος κίνδυνος και γι' αυτό το θέμα του κόστους των μετατροπών νομισμάτων απαιτεί να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια γιατί η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή και ελπίζω ότι από τις τροπολογίες θα προκαλυφθεί μια καλή συνεργασία. Κάποιοι από εσά έχουν εκφράσει επίσης και τις, ε, τη συμφωνία τους για κάποιες ε, χρονικές προθεσμίες πιο φιλόδοξες από αυτές που προτείνονται στην παρούσα φάση. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία λοιπόν. Λοιπόν, διαβάζω το ε, χρονοδιάγραμμα. 14 Σεπτεμβρίου, προθεσμία υπολογής υποβολής επιτροπών, 8 Οκτωβρίου και μετά 5 ε, στην πρώτη ολομέλεια του Νοεμβρίου θα γίνει η ε, ψηφοφορία. Περνάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο αποτελεί σχέδιο έκθεσης για το να συμπεριληφθεί ο Ιταλικός Δήμος Καμπιόνε Ιταλία και τα Ιταλικά Ήδατα της Λίμνης Λουκάνος στην τελωνιακή ε, επικράτεια της Ένωσης και στην ε, εδαφική ε, εφαρμογή της Οδηγίας 2008-118 στο πλαίσιο του κανόνα 5 απλουστευμένης ε, διαδικασίας δεδομένου του υψηλού φόρου εργασίας και της απλής φύσης της πρότασης. Εγώ είμαι εισηγητής εκ μέρους του Προεδρείου. Το κείμενο του σχεδίου έκθεσης δεν ε, προτείνει τροπολογίες της πρότασης της ε, Κομισιόν η οποία σκοπό έχει την τροποποίηση των οδηγιών ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά το με σκοπό μάλλον να συμπεριληφθεί η, ο Ιταλικός Δήμος του Καμπιόνε Τιτάλια και τα ε, της, τα ιταλικά ύδατα της, Λουγκάν, της λίμνης Λουγκάνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία προς το παρόν έχουν αποκλειστεί λόγω γεωγραφικών λόγων όπως η απομόνωση, η μειονεκτική οικονομική θέση, ε, ιστορικά έχει δικαιολογηθεί ο αποκλεισμός από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η Ιταλία θεωρεί ότι αυτός ο αποκλεισμό δεν είναι πλέον απαραίτητος και μετά από Ιταλικό έτοιμο η Κομισιόν πρότεινε οι δύο αυτές περιοχές να περιληφθούν στο, στην τελωνιακή επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην, ε, Ένωση, επικράτεια της Ένωσης όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Παρά τα αυτά η Κομισιόν προτείνει και πάλι ε, ερμηνεύοντας τις επιθυμίες της Ιταλίας να συνεχιστεί ο αποκλεισμό των δύο αυτών περιοχών της εδαφικής εφαρμογής της οδηγίας ε, ΦΠΑ όσον αφορά το, το κοινό σύστημα επιβολής έστω να διατηρηθεί ισότητα μεταξύ των οικονομικών παραγόντων στην Καμπιόνε Ιταλία και στην ε, Ελβετία. Αυτό θα γίνει μέσω έμεσου τοπικού, ε, ε, ε, τοπικού συστήματος έμεσων φόρων. Η πρόταση ζητά απλώς μια επίσημη αλλαγή στην οδηγία ΦΠΑ, από, δηλαδή την μεταφορά των δύο αυτών περιοχών από το σημείο 6,2 στο άρθρο 6,1, το οποίο αφορά τις περιοχές που αποτελούν μέρος της ε, τελωνιακής επικράτειας. Υποστηρίζω, όπως σας είπα, την πρόταση και το σχέδιο έκθεσης ζητώ από το Συμβούλιο να την ε, εγκρίνει ταχύτατα. Έχω δύο μόνο σκιώδεις ε, εισηγητές οι οποίοι παρίστανται και με Πρώτο, τον κύριο Γκίγκολτ. Ε, εκπλήσω Ένα άλλο ιταλικό θέμα. Έχουμε πολλά ιταλικά ζητήματα την, την περίοδο αυτή. Από τις ειδήσεις το πρωί με τις ειδήσεις το βράδυ να είμαστε και στην ΕΚΟΝ. Υποστηρίζουμε σαφώς να συμπεριληφθεί το καμπιόνε. Καμπιόνε, καμπιόνε είναι η σωστή ε, προφορά. Καμπιόνε Ιταλία λοιπόν και τα Ιταλικά ύδατα της Λίνης Λουγκάνος την ε, Τελωνιακή Ένωση. Παρά τα αυτά, όπως και εσείς είπατε πρόεδρε, σημειώνουμε ότι δεν προτείνει η Κομισιόν να συμπεριληφθούν οι δύο αυτές περιοχές και στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΦΠΑ, παρότι η κοινή αναθεώρηση, επανεξέταση των κανόνων του ΦΠΑ θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία. Δεδομένου ότι το Καμπιόνε έχει το μεγαλύτερο καζίνο της Ιταλίας και προτείνω να δείτε όλη τη φωτογραφία του καζίνο, το οποίο στόχευσε μόλις πριν ένα μήνα τον, και ως εκ τούτου ο Δήμος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, διερωτώμαστε αν το, ο Δήμος Καμπιόνε μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ε, φορολογική απάτη συμπεριλαμβανομένης και της απάτη του ΦΠΑ και άρα ε, διερωτώμαστε αν θα πρέπει να μην συμπεριληφθεί στον, στο, στο πεδίο εφαρμογής ΦΠΑ. Αντίθετα, θέλουμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να προτείνει στο Συμβούλιο για να απαλλαγεί από ολόκληρο τον κατάλογο των περιοχών που απαλλάσσονται από το ευρωπαϊκό ΦΠΑ, περιλαμβανομένων και των Channel Islands, όπως ε, προβλέπει το άρθρο 8 της ε, οδηγίας ΦΠΑ. Και αυτό αφορά συγκεκριμένα και τον ε, ανταγωνισμό και στον τομέα των ιδίων πόρων. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Κομισιόν να μας εξηγήσει εν συντομία για ποιο λόγο δεν χρησιμοποίησαν αυτή τη δυνατότητα μέχρι τώρα. Ούτε όταν ε, πρόκειται για το Καμπιόνε, αλλά και στην περίπτωση των άλλων απαλλασσομένων περιοχών. Ευχαριστώ. Δυστυχώς η Κομισιόν δεν παρίσταται, λέει ο Πρόεδρος, όμως θα του ζητήσουμε να στείλουν ε, γραπτή απάντηση στον κύριο Γκίγκολτ. Είναι περίεργο να μην παρίστανται. Είναι ασυνήθιστο. Πρέπει να σημειώσουμε... Όχι, όχι, ο πρόεδρος. Ειλικρινά αυτό επειδή αποφασίστηκε από τους συντονιστές να εφαρμοστεί η απλουστευμένη διαδικασία. Σε αυτό οφείλεται η απουσία της Κομισιόν. Γιατί αρχικά δεν υπήρχε καμία αμφισβήτηση, δεν είχε ζητήσει καμία ε, πολιτική ομάδα κάτι άλλο. Γι' αυτό φυσικά αν υπάρξει αμφισβήτηση τότε εννοείται θα περάσουμε στην κανονική διαδικασία οπότε θα ακολουθήσουμε όλα τα βήματα που περιλαμβάνει η διαδικασία. Τώρα, ολοκληρώσατε, Σβέν, ναι. Επόμενος παρόν ε, σκιώδης είναι ο Μιγγέλ Βιέγκας. Πολύ σύντομα, δεν έχω καμία αντίρρηση από αυτού. Είναι ένα αίτημα του Ιταλικού κράτους. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η ρύθμιση ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και της περιφέρειας. Δεν έχουμε αντίρρηση. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Στο, στη διαδικασία του Catch the Eye θέλει κάποιος το λόγο. Όχι. ως πρώτη διαδικαστική παρατήρηση σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία όπως γνωρίζετε η προθεσμία είναι η 6η Σεπτεμβρίου για την υποβολή αντιρρήσεων αν δεν υπάρχουν λοιπόν ενστάσεις θα περάσουμε άμεσα στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια στην 1η του Οκτωβρίου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 50. Επί της ουσίας, το status quo είναι ότι αυτός ο, ε, χώρος που ανήκει στην Ιταλία ε, απαλλάσσεται από την Τελωνιακή Ένωση και προτείνουμε να συμπεριληφθεί στην Τελωνιακή Ένωση. Θα παραμείνουν τα πράγματα όσο έχουν τώρα, αν δεν κάνουμε τίποτα. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί, θεωρώ ότι είναι θετικό το βήμα αυτό, δηλαδή το να συμπεριλάβουμε αυτά τα εδάφη στην Τελωνιακή Ένωση. Και η πρότασή μας υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα διαβάσουμε βέβαια προσεκτικά και την γραπτή απάντηση της Επιτροπής και θα κρίνουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστώ. Και περνάμε στο επόμενο σημείο και θα αναλάβει την Προεδρία ο Ζήμων. Okay. Liebe Kolleginnen und Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ήδη καθυστερήσει 10 λεπτά και περνάω κατευθείαν στο σημείο 15. Πάλι βάση της απλουστευμένης διαδικασίας, βάση του άρθρου 50. Εδώ έχουμε ένα, ένα σχέδιο έκθεση για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωση όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ιβάνα Μαλετίτς και της δίνω το λόγο για τρία λεπτά και μετά θα δώσω το λόγο στους σιώδεις εισηγητές, δύο λεπτά στον καθένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η, προτινόμενη τροποποίηση του κανονισμού διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωση όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου είναι σημαντική, διότι το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου θα εναρμονιστεί τεχνικά με το νέο σύστημα της οδηγίας για τις γενικές ρυθμίσεις ε, για τους ειδικού φόρους κατανάλωσης που αναδιατυπώνονται. Είναι σημαντικό λοιπόν να είναι εναρμονισμένα τα δύο. Οι νέε ρυθμίσεις στην οδηγία θα απαιτεί την εγγραφή των οικονομικών φορέων που διακινούν προϊόντα βάσει του κεφαλαίου 5 ούτως ώστε να έχουμε αυτοματοποιημένη εποπτεία της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε ένα κράτος μέλος και διακινούνται σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να παραδοθούν για εμπορικούς σκοπούς στο άλλο κράτος μέλος. Για να παρακολουθούμε τις ροές αυτές, τροποποιείται ο κανονισμός και θα περιλαμβάνονται δύο νέες κατηγορίες οικονομικών φορέων διότι χωρίς αυτές τις αλλαγές του Μητρώου δεν θα μπορούσαμε να έχουμε σωστή εποπτεία της διακίνησης. Θα έχουμε λοιπόν τώρα τους ε, πιστοποιημένους αποστολής εγγεγραμμένοι ως αποστολή για υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση και η άλλη κατηγορία είναι οι πιστοποιημένοι παραλήπτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως παραλήπτες για υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση. Το ηλεκτρονικό αρχείο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα του εγγεγραμμένου αποστολέα να αφήνει κενά τα πεδία του προορισμού στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου κατά τη διακίνηση που μέχρι τώρα αυτό ε, ίσχυε για τους εγκεκριμένους αποθηκευτές, σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας. Έχουμε εναρμόνιση λοιπόν ε, του συστήματος αυτού με την οδηγία γενικότερα και μπορούμε να υποστηρίξουμε την πρόταση της Επιτροπής. Δεν χρειάζεται κάποια περαιτέρω τροπολογία και πιστεύω ότι μπορεί βάσει της απλουστευμένης διαδικασίας να γίνει δεκτή η έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ Ιβάνα. Εκ μέρους του ECR, σκιώδης συζητητής, δεν είναι παρόν. Κάποιος άλλος που θα αντικαταστήσει τον σκιώδη εισηγητή δεν βλέπω να είναι στην αίθουσα. Εκ μέρους των φιλελευθέρων να δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Βίρινγκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής και συμφωνώ να προχωρήσουμε βάσει της απλουστευμένης διαδικασίας. Η συνεργασία και τη διοικητική απλούστευση με τη χρήση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ, εφόσον έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ανησυχίες σχετικά με την τήρηση του απορρίτου. Και εφόσον όλα αυτά είναι ε, σύμφωνα με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Ε, οι προτινόμενες αλλαγές θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα για ε, να μπορεί να γίνεται καλύτερα η διακίνηση των προϊόντων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μόλις κολ κάτω, εκ μέρους των Πρασίνων, δεν είναι παρούσα, δεν αντικαθίσταται από κάποιον άλλον. Θέλετε και πάλι το λόγο. Όχι, η συγκήτρια δεν θέλει το λόγο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Σύμφωνα με τον κατάλογό μου δεν έχουμε κάποιο σκιώδη από τους σοσιαλιστές, αλλά πέρνω αν θέλεις το λόγο ευχαρίστως. Μαντίν Τελβό είναι η σκιώδη συζητήτρια και μου ζήτησε να την αντικαταστήσω. Θα ήθελα να το σημειώσει η γραμματεία. Χαίρεται για τις προτάσεις της Επιτροπής, διότι συνάδουν προς τους στόχους μας για την φορολογική πολιτική. Συνεισφέρει αυτή η πρόταση στο να κλείσουμε κάποια παραθυράκια και να αποφεύγουμε την φοροδιαφυγή ενισχύεται η διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερως. Και τέλος, η πρόταση συνεισφέρει στην απλούστευση της διαδικασίας και προωθεί την ψηφιοποίηση, το οποίο είναι θετικό. Η Σκιώδη εισηγήτρια λοιπόν χαιρετίζει το σχέδιο έκθεσης της εισηγήτριας και συμφωνεί να προχωρήσουμε με την απλουστευμένη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Περβάνς. Ζητώ συγγνώμη και πάλι. Στο κατάλογό μου δεν υπήρχε σκιώδης ε, από τους σοσιαλιστές. Επίσης, Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, προθεσμία υποβολή τεραπολογιων Η υποβολή θα γίνει την πρώτη ε, ολομέλεια του Οκτωβρίου. Τώρα, σημείο 16 ήδη οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ εξετάζεται επίσης και μια, ένα σχέδιο γνωμονότησης. Αρμόδια Επιτροπή είναι Μπάντζ, εισηγητής μας είναι ο Ραμόν, έχει το λόγο για 6 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι πρόκειται για μια πρόταση του Συμβουλίου επί τη βάση μιας προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει σαν στόχο την ρύθμιση και τον εξυγχρονισμό του συστήματος ιδίων πόρων. Ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για το σύστημα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόκτηση ιδίων πόρων από τους εθνικούς προϋπολογισμούς είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να ρυθμίσουμε και σε επίπεδο πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ε, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση αλλά είναι και μια πολύ δύσκολη πρόταση. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο και η αίσθησή μας ε, είναι σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο σαν ΕΚΟΝ Η άποψή μας λοιπόν είναι θα έλεγα σας θυμίζω συμβουλευτική ε, και μόνο συμβουλευτική και εδώ το Συμβούλιο είναι σε θέση να προχωρήσει ουσιαστικά μόνο του. Πάντως υπάρχουν δύο τμήματα στην πρόταση. Το πρώτο τμήμα εξυγχρονίζει τους ιδίους πόρους, το παρόν σύστημα και ένα δεύτερο τμήμα ασχολείται με πιθανούς επιπλέον πόρους. Για το πρώτο κομμάτι ουσιαστικά το Συμβούλιο δεν είναι και ιδιαίτερα φιλόδοξο και στην ουσία θέλει να έχει τρία είδη πόρων. Καταρχάς θέλει το λεγόμενο την ενιαία φορολογική βάση επιβολής των επιχειρήσεων και ένα τμήμα πηγαίνει μικρό μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά υπάρχουν τα δικαιώματα έκδοσης, και ένα τρίτο τμήμα είναι οι συνεισφορές τις οποίες μπορεί να κάνουν τα κράτη-μέλη σε σχέση με τα πλαστικά τα οποία ανακυκλώνουν στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Συνεπώς οι τοπολογίες τις οποίες εγώ παρουσιάζω βασίζονται στο ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ περισσότερο φιλόδοξοι σε σχέση με πιθανούς επιπλέον πόρους. Ε, δεν είναι εύκολο βέβαια να το κάνουμε αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προτείνει το Κοινοβούλιο. Ασχολούμε με τέσσερα επιπλέον νομισματικά έσοδα από το ευρωσύστημα. Μιλάμε ουσιαστικά για τα κέρδη της Κεντρικής Τράπεζας που έτσι κι αλλιώς λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των μηχανισμών των επενδυτικών που έχει δημιουργήσει για χώρες με υψηλή ανεργία. Ο, η ίδια η ομάδα εργασίας του κυρίου Μόντι είχε κάνει κάποιες προτάσεις σε σχέση με τους ιδίους πόρους, αλλά δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το έλαβε υπόψη. Δεύτερον, υπάρχει δυνατότητα κάποιων ε, επιπλέον εσόδων από τις συναλλαγές σε ομόλογα μετοχές κτλ. Ε, υποτίθεται ότι για να έχουμε ένα ισορροπημένο προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπονται τέτοιου είδους ε, συγκυριακές, ταμιακές συναλλαγές. Νομίζω ότι αυτή η ιδέα, ούτε και αυτή η ιδέα λαμβάνεται υπόψη. Εγώ νομίζω ότι σαν κοινοβούλιο τουλάχιστον θα έπρεπε να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Και τρίτον, μία ακόμα δυνατότητα, ίσως λίγο πιο μακρινή, η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα επενδυτικό ταμείο, ένα μεγάλο επενδυτικό ταμείο το οποίο να είναι σε θέση να κάνει τις επενδύσεις που χρειάζονται, να δανείζει χρήματα, να δανειοδοτεί με πολύ χαμηλά επιτόκια κτλ. Και τέταρτον κάτι πάλι το οποίο έλεγε ε, η πρόταση Μόντι για τις εισαγωγές ε, από χώρες οι οποίες έχουν υψηλότατα επίπεδα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για να αντισταθμίσουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε περιβαλλοντικό dumping. Νομίζω ότι με τις λεγόμενες ρήτρε Πασρέλ είναι δυνατόν να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε λίγο τις ε, προτάσεις αυτές. Τώρα δεν έχω χρόνο για να σας δώσω περισσότερα στοιχεία, αλλά νομίζω ότι αυτές οι 4-5 ιδέες τις οποίες προσπάθησα να σας εξηγήσω δείχνουν τις απόψεις μου. Σα ευχαριστώ για δύο λεπτά, Ισκιώδης, για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο νέος συντονιστής, τον συγχαίρω γι' αυτό, ο Μάρκους Φέρμπα. Ευχαριστώ, αντικαθιστώ τον Αλένη Λαμασούρ και όταν λέω εγώ δεν μιλάω για μένα αλλά για εκείνον. Λέει λοιπόν ότι καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια πολύ ενδιαφέρουσα και ενδελική εργασία επί του θέματος. Όλοι συμφωνούμε. Το θέμα είναι σημαντικό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Brexit. Ε, μας αναγκάζει να προχωρήσουμε σε καινοτόμους τρόπους για την, για την βιωσιμότητα ε, της Ένωσης και χαίρομαι που μπορώ να συνεργαστώ με τον εισηγητή επ' αυτού. Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του εισηγητή θα ήθελα να εκφράσω δισταγμό όσον αφορά τις διάφορες αποκλήσεις από τις συστάσεις που έχουν διατυπωθεί από την HRGOR, λέει ο μιλητή των ιδίων πόρων. Κυρίως ε, αντιμετωπίζω με σκεπτισμό το θέμα των εσόδων που προέρχονται από του ιδίους πόρους για την ε, χρηματοδότηση την ευρωπαϊκή, ε, τον ευρωπαϊκό τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθεροποίηση ενώ το HG έχει διαφορετική πρόταση. Επίση, όσον αφορά τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κρατικού Ταμείου, European Sovereign Fund, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δούμε πώς θα διαρθρωθεί με τα ε, υφιστάμενα ταμεία όπω ο ΕΦΣΥ. Επίσης το θέμα των, του χρέου, της χρήσης του χρέους και των ομολόγων θα μας απομακρύνουν από το σημαντικό θέμα των ιδίων πόρων και θα χαθούμε στη συζήτηση. Όσον αφορά τις επιστροφές, θεωρώ ότι ο εισηγητής και εγώ βρισκόμαστε σε συμφωνία και θα ήθελα και εγώ να συνεισφέρω στη διατύπωση αυτής της θέσης. Θα πρέπει να γίνει διόρθωση το ταχύτερο δυνατό, κυρίως δεδομένου ότι η αναχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ε, Ένωση εκμηδενίζει το αρχικό νόημα. Επίσης θα ήθελα να συμφωνήσω με τον εισηγητή που ζητά από το Συμβούλιο ε, την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μια ε, εξαιρετική νομική διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε γρήγορα τις διαπραγματεύσεις αυτές. Προσβλέπω σε περαιτέρω συζήτηση των θεμάτων αυτών με τον εισηγητή. Αυτά ήθελε να πει ο Άλαν. E ευχαριστώ πολύ για το ECR. Ο Μπραντ Λούκε, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης. Ε, έχω δύο παρατηρήσεις ε, και μετά από αυτά που ακούσαμε εκ μέρους του ΕΛΑ, επίσης θέλω να το πω. Έχουμε το σύστημα των εθνικών τραπεζών και τα κράτη-μέλη μέσω των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, θα πρέπει να λαμβάνουν ε, τις ε, αποφάσεις. Μέχρι τώρα δεν είχαμε άμεση πρόσβαση στα κέρδη της Κεντρικής Τράπεζας. Και αυτό το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο επίσης είναι ένα καινούριο στοιχείο έχουμε την πρόταση της Επιτροπής, που δεν τη θεωρώ ιδιαίτερα καλή, και θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Η Επιτροπή ε, δεν αποδεικνύει ότι το παρόν σύστημα είναι κακό. Ε, το επιχείρημα σχετικά με το ΑΕΠ ως ιδιοπόρο δεν είναι επαρκές γίνεται όλο και πιο ε, ε, πολύπλοκο το σύστημα και δημιουργεί ε, fake news. Με το καινούριο σύστημα δεν βλέπουμε ποιο είναι το πρόβλημα με τον ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη με την διάβρωση της βάσης του ΦΠΑ. και επομένως ε, πώς μειώνεται η βάση των ιδίων πόρων της κοινότητας. Ε, η νέα πρόταση ε, για τον φορετεριών δεν περιλαμβάνει όλες τις, όλα τα κράτη-μέλη και δεν είναι σαφές πώς θα γίνει ίδιος πόρος που θα επιβάλλεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορούμε να, θεωρήσουμε ότι καταβάλλεται από όλα τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τις ε, εκπομπές, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, δεν έχει συζητηθεί αρκετά, και τα απορρίμματα πλαστικών ε, είναι κάτι όπου βλέπω ότι προσπαθούμε να βρούμε πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει καταρχήν να εφαρμόσουμε την αρχή του ότι ο ρηπαίνων ε, πληρώνει. Γιατί θα πρέπει ε, μέσω του συστήματος εκπομπών ε, να φροντίσουμε να επιβαρύνονται οικονομικά αυτοί οι οποίοι ρηπαίνουν περισσότερο. Ευχαριστούμε κύριε Λούκε. Η κυρία Βίρινκα, εκ μέρους του Άλντε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή και για τις προτάσεις που μας κάνατε. Είναι πολύ φιλόδοξη η πρόταση αυτή, ίσως και υπερβολικά φιλόδοξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως δεν μπορεί να λειτουργήσει ε, σωστά και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών της χωρίς τους κατάλληλους πόρους. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε μεγαλύτερη ε, δημοσιονομική ανεξαρτησία. Και είμαι πεπισμένη ότι αυτό θα είναι προς όφελος και των κρατών μελών, διότι ήδη πόρη σημαίνει και ανάληψη των ευθυνών μας. Έχω τις εξής παρατηρήσεις. Ο εισηγητή ανέφερε ένα ευρωπαϊκό ταμείο. Τι είναι αυτό το European Sovereign Fund και ποιος θα είναι ο ρόλος του. Δεύτερον, όσον αφορά τα ευρωομόλογα, ο επιμερισμένος κίνδυνος σημαίνει χαμηλό κίνδυνο όλοι θα πρέπει να έχουν συμπεφωνημένους κανόνες και φοβούμαι ότι η τρέχουσα πολιτική προτεραιότητα είναι διαφορετική. Και τρίτον, δεν θα ήθελα να συμφωνήσω ε, με αυτό το οποίο προτείνονται για τα έσοδα. Οι πόροι θα πρέπει να είναι πόροι ευθυγραμμισμένοι με την έκθεση Μόντι και να μην επιβάλλουμε νέους φόρους στους πολίτες μας. Και ε, θα επιμείνω στο ότι οι δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβαδίζουν με τα έσοδά τη. Ο δανεισμό από τι διεθνεί αγορέ μπορεί ε, να θέσει σε κίνδυνο αυτή η γενική αρχή. Ευχαριστώ πολύ και θα τα συνεχίσουμε να τα συζητάμε κατά τι επόμενε εβδομάδε. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου των Πρασίνων, κύριε Σουρτασούν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης και συμφωνώ με πολλές από τις προτάσεις που έκανε και συμφωνούμε με την μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων. Το 80% ε, χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους ε, και αυτό δημιουργεί συζητήσεις για τα θέματα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι διαφανής ε, και δίκαιος ο τωρινός διακανονισμός. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που θα είναι δίκαιο για όλες τις περιφέρειες και θα έχει και μια ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική. Οι πράσινοι υποστηρίζουν την πρόταση να έχουμε τρεις νέους ίδιους πόρους συνεισφορά από την ΕΚΤ, από το σύστημα εκπομπών και τον φόρο από τα πλαστικά. Επί χρόνια επιμένουμε και χαιρόμαστε που η Επιτροπή ακολουθεί αυτές τις προτάσεις. Θέλουμε να μειώσουμε τη συνεισφορά εκ μέρους του ΑΕΠ και να έχουμε ένα προϋπολογισμό που θα χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και όχι από εθνικές συνεισφορές. Και υποστηρίζουμε την πρόταση για τροποποίηση των ε, ίδιων πόρων ε, σύμφωνα με τις ε, απόψεις που έχει εκφράσει το Κοινοβούλιο. Οι επιστροφές τέλος δεν είναι μια έννοια που έχει νόημα και μπορεί να χρειαστεί μία πενταετής περίοδος για τη σταδιακή εξάλληψη αυτού του συστήματος των επιστροφών. Γενικά συμφωνούμε με το σχέδιο έκθεσης ε, του εισηγητού. Περιμένουμε περαιτέρω τροπολογίες γιατί ε, για να είμαστε αρκετά φιλόδοξοι θα πρέπει να κάνουμε τις κατάλληλες τροποποίησεις στο κείμενο αυτό και στην πρόταση της Επιτροπής και στο πλαίσιο των συζητήσεών μας θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ποια είναι η καλύτερη μέθοδος ένας φόρος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ένας φόρος επί των αεροπορικών μεταφορών, των ε, τηλεπικοινωνιών είναι φόροι που θα πρέπει να συζητηθούν. Θέλουμε ε, να ε, βελτιωθεί το σύστημα και το ανώτατο όριο για τους ιδίους πόρους και τέλος δεν θα πρέπει να υπάρχει φορολογία χωρίς εκπροσώπηση και ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την εκπροσώπηση των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα υποβάλουμε μια σχετική τροπολογία προσωμιάζει με την τροπολογία 41 του εισηγητού. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στις συζητήσεις μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ε, τον συνάδελφο Χαουρέγγι, για το σχέδιο γνωμοδότης που παρουσίασε και συμφωνώ με τη βασική θέση που μας παρουσίασε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι πιο φιλόδοξο στην προσέγγιση του θέματος των ιδίων πόρων. Και διαφωνώντας με αρκετούς σκιώδεις ηγητές που προηγήθηκαν, που ανήκουν στον συντηρητικό πολιτικό χώρο, θα έλεγα ότι οφείλουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είμαστε πιο φιλόδοξοι από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο, με βάση και τις απόψεις που το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αντίθετο με την προσέγγιση που λέει ότι χρειάζεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός διαρκώς να συρρυκνώνεται και ότι το Brexit είναι μια ευκαιρία για να συρρυκνωθεί κι άλλο. Και επειδή αυτή η πολιετής διαμάχη ανάμεσα στα κράτη-μέλη καθαρούς εισφορείς και τα κράτη-μέλη καθαρούς δότες, net contributors εναντίον net receivers και vice versa, οδηγεί σε αδιέξοδα και σε καθυστερήσεις και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 πρέπει να προετοιμαστεί εν ώψη και του Brexit, πρέπει εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο να μην επιτρέψουμε να πεταχθούν στα σκουπίδια οι προτάσεις της Επιτροπής Μόντι, αλλά να προτείνουμε και άλλους ίδιους πόρους. Επομένως, με αυτό το πνεύμα της αύξησης των ιδίων πόρων, που θα αυξήσουν και το ποσοστό της συμβολής των ιδίων πόρων με αντίστοιχη μείωση των εθνικών συμβολών των κρατών μελών, θα κινηθούμε σε συνεργασία με τον εισηγήτη και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές, στη φάση της συζήτησης των συνεδριάσεων και της διαμόρφωσης και διατύπωσης τροπολογιών. Εγώ όμως θέλω να στηριχτούμε κάποια στιγμή και στην κοινή λογική είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χωρίς τους κατάλληλους πόρους. Είναι δυνατόν να αφήσουμε την ε, έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων να μεγαλώνει και τις ανισότητες περιφερειακές και κοινωνικές να μεγαλώνουν και εμείς να λέμε προς Θεού μην αυξήσουμε τους ίδιους πόρους. Όσοι το κάνουν αυτό εργάζονται για τους ακροδεξιούς λαϊκιστές που θέλουν τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να λέμε θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε φιλοευρωπαϊστές, θέλουμε κοινωνική πολιτική, θέλουμε ε, επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, θέλουμε αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θέλουμε περισσότερη κοινωνική συνοχή, αλλά όταν ερχόμαστε στη στιγμή που πρέπει αυτά να χρηματοδοτηθούν, εκεί να υπάρχει ένα όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Κανείς εκπρόσωπος από την ΕΝΕΦ. Δίνω το λόγο και πάλι στον εισηγητή για ένα λεπτό. Ένα λεπτό μόνο, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για όλα τα σχόλια. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές Γνωρίζω ότι δεν συμφωνούμε όλοι ε, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης και ξέρω ότι οι προτάσεις μου προσπαθούν να δώσουν περισσότερες δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, αποσκοπούν στο να εξαρτώμεθα λιγότερο από τις εθνικές συνεισφορές. Αυτό είναι μια πολιτική φιλοσοφία. Είναι το πνεύμα της ομάδας μου. Και αυτό ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει αύξηση των ιδίων πόρων. Θα θέλαμε στα επόμενα χρόνια από 8 να περάσουμε στο 18%. Για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε, χρειάζονται κάποιες δημοσιονομικές επιλογές. Ποια είναι λοιπόν η φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει η κοινή βάση φορολογίας εταιριών, υπάρχει ο ΦΠΑ. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι η εναρμόνιση. Διαφορετικά θα ισχύσει αθέμητος ανταγωνισμός. Σε ορισμένες χώρες όντως υπάρξει, υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός και την φορολογία των εταιριών, είναι σαφές ότι υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμός και ο κύριος Ζήμων γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι απαραίτητο να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ενιαία αγορά. Αυτή η φιλοσοφία βρίσκεται πίσω από την ε, πρότασή μας. Θα πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένες πολιτικές. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο στην ουσία εμένουν στην ανακύκλωση των πλακτικών. Υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, δεν έχουν προχωρήσει πολύ και θα χάσουν λίγο περισσότερο. Γι' αυτό εγώ θυμίζω ότι ο κύριος Μόντι είχε προτείνει την δυνατότητα στα πλαίσια των δικαιωμάτων ε, εκπομπών να υπάρχει ένα τμήμα το οποίο να καταλήγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς προσπαθούμε να αποτρέψουμε λοιπόν το περιβαλλοντικό dumping ε, από χώρες δηλαδή που εισάγονται προϊόντα από χώρες οι οποίες έχουν υψηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και εδώ υπάρχουν κάποιες διαφορές που μπορεί να έχουν ε, και φιλοσοφική θα έλεγα διάσταση. Εγώ πάντως πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να είναι πάρα πολύ φιλόδοξος σε σχέση με τους ιδίους πόρους έτσι ώστε να αυξήσει τον κατάλογο των ιδίων πόρων. Τα οικονομικά έσοδα του ευρωσυστήματος χρησιμοποιούνται ήδη ουσιαστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει φτιάξει έναν κανονισμό όπου υπάρχουν επιστροφές και αντισταθμίσεις για ορισμένες χώρες στα πλαίσια των κεντρικών τους τραπεζών. Συνεπώς λοιπόν δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε αυτά. Σα ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε διότι έχω μιλήσει περισσότερο αλλά θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε την μέγιστη δυνατή συνένεση εκεί όπου υπάρχει δυνατότητα. Αν δεν υπάρχει τώρα θα δούμε. Ευχαριστώ Ραμόν. Λοιπόν, 4 Σεπτεμβρίου τροπολογίες θα μελετήσουμε θα μελετηθούν τέλος Οκτωβρίου και στις 8 ή 9 Οκτωβρίου θα γίνει η 9 οκτωβριου θα γινει ψηφοφορια για την έκθεση. Επόμενο θέμα, θέμα 17, η προστασία ατόμων που ε, καταγγέλουν παραβιάσεις του ενωτικού δικαίου. Έχουμε μέλλον, ε, και ερευνητικές επιτροπές για τα έγγραφα του Παναμά και άλλες. Ε, είναι πολύ σημαντικό άρα το θέμα. Ο εισηγητής είναι ο Μικέλ Βιέγας. Η επιτροπή μας είναι συνδεδεμένη επιτροπή με βάση τον, τον κανόνα 54 με αποκλειστική αρμοδιότητα σε θέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, φορολογίας και ανταγωνισμού. Μικέλ, έχει το λόγο. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή πρέπει να τύχει ευρεία συνένεση. Όλοι αντιλαμβάνεστε, είμαι βέβαιος, την μεγάλη σημασία του θέματος. Άρα είμαι αισιόδοξο. Θα μπορέσουμε να έχουμε ένα ενοποιημένο κείμενο που θα εκφράζει όλες μας τις επιθυμίες. Η έκθεση ενώπιόν σας Είναι έκθεση την οποία προσπάθησα να βελτιώσω. Έκανα αλλαγές, όμως ουσιαστικά θέλησα να ανακεφαλαιώσω αυτό που ήθελα να, βελτιώ, να κάνω, δηλαδή να βελτιώσω τον ορισμό, να διευρύνω το πεδίο εφαρμογής της ίδιας της οδηγίας Υπάρχει η εντύπωση ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί καν να λειτουργήσει. Ότι δηλαδή θα πρέπει οι ίδιες οι κυβερνήσεις να ε, εξασφαλίσουν το σωστό έλεγχο και την επίβλεψη. Για μας είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι θα βάλουμε υπερβολικά μεγάλη ευθύνη ε, στους καταγγέλλοντες έναντι της κυβέρνησης. Δεν θέλω η βασική ιδέα της έκθεσης τελικά να είναι ότι τα κράτη μπορούν να απαλλαγούν από τις ευθύνες τους ε, του σωστού ελέγχου της έρευνας και της επιθεώρησης. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα στην έκθεση. Θα επικεντρωθώ σε δύο. Πρέπει να αγγιηθούμε την ανωνυμία πρώτον. Πρέπει να στηριχθούμε στις εμπειρίες μας και τις επαφές μας με καταγγέλλοντες στο παρελθόν. Πρέπει να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς όταν αναφέρουν προβλήματα Θεωρώ ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε γιατί επιθυμούν την ανωνυμία. Πρέπει να είναι σαφές αυτό. Υπάρχει και η γενικότερη ιδέα στην πρόταση αυτή ότι θα πρέπει τα η εξωτερική διαβλή να, να είναι ε, υποδέστερη των εσωτερικών. Δεν το θεωρώ απαραίτητο. Αυτός που κάνει την καταγγελία πρώτα πρέπει να περάσει από μια εσωτερική αναφορά εντός της επιχείρησης και όταν έχουν εξαντληθεί όλες αυτές οι δυνατότητες μπορεί να κινηθεί χρησιμοποιώντας εξωτερικούς διάβλους. Αυτό είναι κάπως υπερβολικό πιστεύω γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία των ε, καταγγελιών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Ελπίζω λοιπόν ότι θα γίνει μια ουσιαστική συζήτηση που θα βελτιώσει την πρόταση της Επιτροπής, η οποία και αυτή αποτελεί ένα βήμα πρόοδου, αλλά αφορά ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί σωστά. Υπάρχουν και άλλα ε, θέματα με τα οποία, τα οποία μπορούμε να προσθέσουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Μιγγέλ. Ο Μπένερ Λάγκεν δεν είναι παρόν. Τον αντικαθιστά κάποιος. Δεν τον αντικαθιστά κάποιος. Ο κύριος Καφούντε επίσης δεν είναι παρόν. Ο Λελόντιξον. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω εκ μέρους του κυρίου Καφούντε. Η ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής. Είναι μια πρόταση που έχει ενισχυθεί και βελτιώθηκε από τον εισηγητή της Επιτροπής Γιούρη με σημαντικές δικλίδες ασφαλείας και προειδοποιήσεις για παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρχει καλύτερη προστασία ε, του απορρίτου για τους καταγγέλτες και προστασία ε, της προσωπικής τους ασφάλειας. Εφαρμόζοντας τις διατάξεις αυτές ε, ελάχιστον μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα ενιαίο και συνεπές πλαίσιο για την προστασία των καταγγελτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει η δυνατότητα των κρατών μελών να θεσμοθετήσουν ισχυρότερη ακόμη προστασία, αλλά το τωρινό πλαίσιο είναι κάτι το οποίο εδώ και χρόνια ήταν απαραίτητο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει σε μια τέτοια πρόταση όπως αυτή που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας. Είναι ένα σημαντικό βήμα πρόοδου και μετά τη δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή μας και η Ειδική Επιτροπή Διερεύνησης ε, Οικονομικών ε, Εγκλημάτων ε, έχουν, έχει καταβάλει επίσης αντίστοιχες προσπάθειες. Θέλουμε να διασφαλίσουμε καλύτερη προστασία για τους καταγγέλτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα έγγραφα του Παναμά, η ε, υπόθεση ε, Paradise, τα Lux Leaks, ε, τα σκάνδαλα για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ναι, είναι σκάνδαλα τα οποία είχαν άμεσα σχέση με την δράση κάποιων καταγγελτών. Τα διεθνή οι διεθνείς προσπάθειες φοροδιαφυγής και ξεπλήματος χρημάτων θα είχαν συνεχιστεί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αν δεν υπήρχαν ε, οι καταγγέλτες. Θα πρέπει να διδαχθούμε από ε, όσα έχουν αποκαλυφθεί στα πλαίσια των υποθέσεων που έχουν συζητηθεί και με βάση των εργασιών των Επιτροπών ΤΑΞ και ΤΑΞ 2 και πάνω και τη συνεχιζόμενη εργασία την ΤΑΚΣ 3 θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Οι καταγγέλτες ε, που ε, κάνουν το θαραλέο βήμα σε περιπτώσεις πολυεθνικών εταιριών πολύ συχνά υπόκεινται σε ποινικέ κυρώσεις. Ενώ πολλές εταιρείες που έκαναν τα οικονομικά εγκλήματα πολλές φορές ε, έχουν διαφύγει πραγματικής τιμωρίας. Και γνωρίζουμε ε, ότι ε, πολλοί δυνητικοί καταγγέλτες σε πολυεθνικές εταιρείες και διεθνείς θεσμούς φοβούνται να κάνουν το βήμα και να κάνουν μια αποκάλυψη. μπορεί να υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπου υπάρχουν προβλήματα και εντός μιας χώρας και διασυνοριακά. Κάποιες αρχές δεν θέλουν να καταγγείλουν άλλες αρχές ή μπορεί οι αρχές κρατών μελών ε, να καθυστερούν και να μην δρουν άμεσα μετά από την ενημέρωση από τους καταγγέλτες. Σε άλλες περιπτώσεις, τα μέτρα που λαμβάνουν ε, μπορεί να μην είναι μέτρα συνεργασίας, αλλά η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών να καταλήγει σε αρνητικά αποτελέσματα. Ε, λόγω της έλλειψης σωστών μέτρων συντονισμού. Γι' αυτό χρειάζονται μέτρα διευκόλυνσης των καταγγελτών σε περιπτώσεις ε, διασυνοριακών υποθέσεων. Η ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής και του εισηγητού και θέλουμε να ενισχυθούν οι προτάσεις ιδίως για την περίπτωση των καταγγελτών σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στη διεθνή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ όλοι. Ρόμπερτ Σίλε για το ECR που δεν είναι παρόν, που εκπροσωπείται από κάποιον. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Μιουέλ Βιέγας για μια εξαιρετική έκθεση, σημαντική για την πολιτική μας ομάδα. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των καταγγελόντων που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Πρέπει λοιπόν να τους προστατεύσουμε όσους ε, καταγγέλουν την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου πρέπει να τους ε, προστατεύσουμε από αντίμετρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες δυνατές πρακτικές Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει αναφορά στην έκθεση αυτή στο hacking και στο κυβερνοέγκλημα, όπως επίσης και στην, στις τρομοκρατικές δράσεις μέσω διαδικτύου, την λεγόμενη κυβερνοτρομοκρατία. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πολύ του συμπολίτε μας. Τον Ιούλιο είχαμε πάει στις Ηνωμένε Πολιτείε και βασική ανησυχία ήταν οι κυβερνοεπιθέσεις, περισσότερο από το οικονομικό έγκλημα. Είδαμε ότι χρησιμοποιούν πολλά μέσα και πολλές πολιτικές για να προστατευθούν από, τις κυβέρνο από το κυβερνοέγκλημα, από τις επιθέσεις σε επίπεδο διαδικτύου να μην ξεχνάμε ότι οι νέες τεχνολογίες δυστυχώς εκτίθενται σε πάρα πολλές απειλές και μιλάμε για παραβιάσεις του, του κοινοτικού δικαίου, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ότι υπάρχουν πολλές παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου σε σχέση με την μεταφορά και την εφαρμογή των κοινοτικών αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ξεκινά σχεδόν χίλιες προσφυγές επί παραβάση. Να σας θυμίσω ότι εδώ ο Μάριο Ντράγκη τον Νοέμβριο υπέστη πάρα πολλές επιθέσεις και ταυτόχρονα κατηγόρησε ε, τα κράτη-μέλη ότι ε, δεν έχουν εφαρμόσει σωστά το κοινωνικό δίκαιο. Είπε λοιπόν ότι η έλλειψη εφαρμογής της οδηγίας για καθυστερημένες πληρωμές οδήγησε ε, σε πάρα πολλές κρίσεις όπως αυτή των κόκκινων δανείων κτλ. Συνεπώς λοιπόν μιλάμε για πάρα πολλά θέματα στα οποία τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να εφαρμόσουν την κοινοτική νομοθεσία με πολύ πιο γρήγορο και σωστό τρόπο. Ευχαριστώ Ραμόν. Δεν έχω κανέναν από την ΚΟΕ FTDNF. Να σας ενημερώσω για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών 4 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Και οι τροπολογίες πρέπει να σας ενημερώσω ότι πρέπει να υποβάλλονται μόνο στα αγγλικά. Γιατί η Επιτροπή Γιούρι θα πρέπει να ψηφίσει τον ε, Οκτώβριο. Δεν ξέρω αν είναι ε, θεμητό και νόμιμο αυτό. Γιατί ο καθένας έχει δικαίωμα να υποβάλει τροπολογία στη μητρική του γλώσσα. Εξέταση των τροπολογιών 24 Σεπτεμβρίου, ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ 24 Σεπτεμβρίου την ίδια μέρα και ψηφοφορία στη Γιούρη 10 Οκτωβρίου. Επειδή είναι πολύ νωρίς η ψηφοφορία, γι' αυτό οι τροπολογίες μπορούν να υποβάλλονται μόνο στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ και περνάμε στο σημείο 18 της ημερήσιας διάταξης, διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διαιρέσεις. Πάλι η Επιτροπή Γιούρη είναι η αρμόδια επιτροπή και ο εισηγητής είναι ο Λούντιξον που του δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρέπει ε, να διευκολύνουμε την κινητικότητα των επιχειρήσεων διασυνοριακά στην ενιαία αγορά ε, και ταυτόχρονα να έχουμε και επαρκή προστασία για την ενιαία αγορά. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα διασφάλισης για να αποφεύγεται οποιαδήποτε κατάχρηση και οποιασδήποτε μεθοδευμένες ε, αλλαγές που μπορεί να καταλήγουν σε κοινωνικό ή φορολογικό dumping. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντική και στην δική μου έκθεση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Οίκων προσπαθώ να εξετάσω την πρόταση της Επιτροπής δεν ε, μπαίνω σε θέματα ε, διαβούλευση με του εργαζομένου, γιατί δεν είναι αντικείμενο τη Επιτροπή μα. Η πρόταση χρειάζεται κάποιε διευκρινήσει και θα πρέπει να φροντίσουμε τα μέτρα διασφάλιση να μπορούν να εφαρμόζονται πλήρω και να μην ε, παραμένει ανοιχτό κανένα παραθυράκι. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει πεδίο ε, παράβασης της φορολογικής νομοθεσίας. Προτείνω να μπει ένας ορισμός ε, που θα καθορίζει τι είναι οι τεχνητές μεθοδεύσεις. Αν δεν υπάρχει σαφής ορισμός, τα κράτη-μέλη ενδέχεται να ερμηνεύουν τους κανόνες με τρόπο που δεν ε, θα είναι κοινός για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν θέλουμε να δημιουργούνται περισσότερες εικονικές εταιρείε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αποτρέψουμε. Επίσης, θέλουμε να επεκταθεί η έννοια των τεχνητών μεθοδεύσεων και να καλύπτει και τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Ε, ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα πιθανά κενά θα καλύπτονται και θα επιτυχάνεται η μέγιστη δυνατή σαφήνεια. Σχετικά με τις τεχνητές μεθοδεύσεις, θα πρέπει να υπάρχει μια πραγματική οικονομική σύνδεση με το κράτος καταχώρησης για να μην γίνεται κατάχρηση της ελευθερίας εγκατάστασης, ιδίως όσον αφορά την φοροαποφυγή. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει και την εξέταση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα πρέπει να γίνεται από μία δημόσια αρχή. Και γι' αυτό έχω υποβάλει και μια τροπολογία. Στην πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπεται κάποια δυνατότητα εκ των υστέρων παρακολούθησης και επιβολής. Αυτό είναι σημαντικό διότι μπορεί να είναι δύσκολη η εκ των προτέρων ανακάλυψη τεχνητών μεθοδεύσεων και γι' αυτό προτείνω μια τροπολογία που εισάγει την έννοια της εκ των υστέρων παρακολούθησης για τις διασυνοριακές μετατροπές όταν δεν πληρούνται οι απαιτήσει. Τέλος, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι σωστό να συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση οι διασυνοριακές διασπάσεις μόνο ένα περιορισμένο εύρος διασπάσεων ε, καλύπτεται. Η διάσπαση μιας εταιρείας σε δύο ή περισσότερες νεοσυσταθήσεις επιχειρήσεις και υπάρχουν αμφιβολίες για το αν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι διασπάσεις. Ίσως καλύτερα να διαγραφεί αυτό το μέρος της πρότασης. Προσβλέπω στις συζητήσεις που θα έχουμε κατά τις επόμενες εβδομάδες με τρόπο ευέλικτο και ελπίζω ότι και οι συνάδελφοι θα συνεργαστούν με ευελιξία για να βρούμε κοινέ λύσεις που θα τύχουν ευρεία υποστήριξη Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ όλε. Άννε Ζάντερς ε, εκπροσωπεί τον ε, κύριο Σβάμπ. Ευχαριστώ συνάδελφοι να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του ΣΒΑΜΠ που δεν μπορεί να είναι ε, μαζί μας σήμερα γι' αυτό θα διαβάσω το κείμενό του. Ο κύριος Σβάμπ λοιπόν δέχεται θετικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι καιρός έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να περιλάβει το κατάλληλο πλαίσιο το οποίο θα καταστήσει πιο εύκολο οι επιχειρήσεις να συγχωνεύονται, να χωρίζονται στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς. Είναι βασικό όμως ένα τέτοιο πλαίσιο να είναι συνεκτικό και συμβατό με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδιαίτερα μετά από την υιοθέτηση της οδηγίας αυτής, οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε χειρότερη θέση σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης όπως την ερμηνεύει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό δυστυχώς δεν διασφαλίζεται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η, Ευρωπαϊκή, η πρόταση λοιπόν του κυρίου Σβάμπ θεωρεί ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης. Ο κύριος Σβάμπ πιστεύει ότι τα, τα προτινόμενα κείμενα 86C και 160D σχετικά με τις συνθήκες ε, για τις διαιρέσεις και συγχωνεύσεις τις διασυνοριακές είναι αντίθετες με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέγουν ότι ε, είναι δυσανάλογη και προκατηλημένη η θεώρηση ύπαρξης ε, καταχρήσης. Συνεπώς, η καταλληλότητα καταπολέμησης ή αντιμετώπισης αδικαιολόγητων και ατεκμηρίωτων ειδικού τύπου φορολογικών ρυθμίσεων δεν αντιμετωπίζεται με τον σωστό τρόπο. Ο σκιώδης εισηγητής λοιπόν του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος απορρίπτει τις προτάσεις αυτές. Η λύση την οποία προτείνει ο κύριος Σβάμπ δυστυχώς πάλι ή μάλλον οι προτάσεις του εισηγητή δεν καλύπτουν τις ανησυχίες του κυρίου Σφαμπ. Ο κύριος ε, ο Σκιώδης πιστεύει ότι οι προτάσεις που γίνονται για τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες είναι υπερβολικές. η εξέταση αυτών των ρυθμίσεων από ανεξάρτητους ε, εμπειρογνώμονες είναι κάτι το οποίο είναι συζητήσιμο. Πόσο μάλλον που εδώ, όπως και σε, άλλες, ε, σε άλλα σημεία της πρότασης, οι ρυθμίσεις ε, για μη υπαρκτό λόγο αποκλίνουν από τους ισχύοντες κανόνες για τις συγχωνεύσεις. Ο κύριος Φαμπ λοιπόν με τις δικές του τροπολογίες ε, θα προσπαθήσει να συνεργαστεί περισσότερο με τους υπόλοιπους. Για το ECR έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κύριε Σιγητά, η ομάδα μου θα στηρίξει τις περισσότερες από τις τροπολογίες σας γιατί έχουν σαν στόχο την καταπολέμηση των απατών στον τομέα της φορολογίας. Επίσης είναι ικανοποιητικός και ο ορισμός που δίνετε εσείς για τις λεγόμενες τεχνητές δομές και ρυθμίσεις το ECR έχει όμως ορισμένες επιφυλάξεις σε σχέση με κάποια άλλα σημεία. Πρώτον, ε, το θέμα της διαίρεσης των επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να μείνει εκτός οδηγίας. Δεύτερον, για τις κυρώσεις. Υπάρχει ένα νέο άρθρο. Νομίζουμε ότι οι προβλέψεις αυτές δεν είναι απαραίτητες. Ακόμα και τώρα τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν κυρώσεις για παράνομες συμπεριφορές. Δεν χρειάζονται λοιπόν επικαλύψεις. Τώρα, σχετικά με την λήψη υπόψη των συμφερόντων των υπαλλήλων και των εργαζομένων, Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με, το ίδιο πρόβλημα. Έχω και κάποια άλλα σχόλια σε σχέση με το πώς ε, η ιδέα των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να λειτουργήσει εκεί όπου γίνεται αναφορά για διασυνοριακές μορφές συνεργασίας, αλλά δεν είναι η συζήτηση τωρινή. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσουμε να εξετάζουμε τα θέματα αυτά στο μέλλον. Και ελπίζουμε ε, να συνεχιστεί η προσπάθεια. Υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεργασίας ανάμεσα στις διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ Σταν ο για την Άλντε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, τον αγαπητό Όλε Λούντβικσον για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς και της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγγνώμη, και της εσωτερικής αγοράς υπάρχει δυνατότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εγκαθίστανται στο σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες φύγονται από τα εθνικά και πολυδιασπασμένα νομικά εθνικά πλαίσια στον τομέα των αγορών, ε, ε, διαχωρισμών επιχειρήσεων και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα η εκ νέου οργάνωση μέσω της ψηφιοποίησης των διασύνοριακών συναλλαγών είναι κάτι που θα επιτρέψει τη μείωση του κόστους για τις μικρομεσαίες απαιτείται να υπάρχει ένα συνεκτικό διεθνές πλαίσιο έτσι ώστε να δίδονται κίνητρα στις επιχειρήσεις για διασυνοριακές δραστηριότητες. Ο εισηγητής στέκεται και στα θέματα ε, της εργασίας και δεν είναι λάθος αυτό, αλλά αυτό θα πρέπει να ισορροπηθεί με μεγαλύτερη προσοχή των αγορών και των φορολογικών ρυθμίσεων. Πιστεύουμε επίσης ότι είναι πολύ καλή ιδέα ή ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμων για την αξιολόγηση των συναλλαγών αυτών. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσουμε από κοινού να καταλήξουμε σε μια συνένεση και σε μια τελική πρόταση. Ευχαριστώ πολύ, Ραμόν. Εκ μέρου των Πρασίνων δεν έχουμε κάποιον. Ε, νομίζω ο Σβέν Γκίγκολ θα λάβει το λόγο εκ μέρου των Πρασίνων για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, θέλω να τονίσω ότι η πρόταση της Επιτροπής έχει μια διπλή γλώσσα. Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προσπαθεί αφενός μεν να περιορίσει τις ζημιές από την, τις επιπτώσεις της απόφασης του δικαστηρίου, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να θέτουν κάποια όρια ε, στα θέματα αυτού του ανταγωνισμού. Από την άλλη πλευρά, θέλει να αυξήσει τον ανταγωνισμό μέσα στα κράτη-μέλη για το πού θα εγκαθίστανται οι επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο τα κάνει τις επιχειρήσεις ε, να μεταφέρουν την έδρα τους. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός για την εγκατάσταση ε, των εταιριών αλλά το σημαντικό είναι ότι έχουν υποχρεώσεις οι εταιρείες ε, στο, σημείο, στο γεωγραφικό σημείο στο οποίο είναι παρούσες. Και γι' αυτό ε, θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα τι σημαίνει ε, τεχνητές μεθοδεύσεις. Και έχει δίκιο η εισηγητής, να μην αφήσουμε τα κράτη-μέλη ε, να αυτοσχεδιάσουν, οπότε ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι αθέμητος, αλλά θα πρέπει να ανταγωνίζονται οι εταιρείε μεταξύ τους και όχι τα κράτη-μέλη μεταξύ τους με κίνητρα για τις επιχειρήσεις ή για το εργατικό δίκαιο ώστε να προσελκύουν εταιρείε. Ας βοηθήσουμε να επικρατήσει η ειρήνη στην εσωτερική αγορά. Να ενισχύσουμε λοιπόν τη διατύπωση στο σημείο που αναφέρονται οι τεχνητές μεθοδεύσεις και επίσης οι διατάξεις που αφορούν τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα θα πρέπει να διαγραφούν και θέλουμε περισσότερους κανόνες για τη διαφάνεια για να επανέλθουν τα πράγματα στο σωστό δρόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Σβέν. Μάρτιν, εκ μέρους της Ευχαριστώ πολύ και πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει άμεση σχέση με το δικαίωμα εγκατάστασης των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα και για τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις. Θέλουμε και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εταιριών και να τηρούνται οι διατάξεις ε, ε, για το θεμητό ανταγωνισμό στα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια πρόταση για διαγραφή του κεφαλαίου 4. Συμφωνεί η ομάδα μου με τη διαγραφή του κεφαλαίου 4, διότι και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος ε, να γίνει κατάχρηση της δυνατότητας που παρέχει η Επιτροπή και θα μπορούν οι επιχειρήσεις ε, να παρακάμπτουν αυτή τη διαδικασία. Συμφωνούμε με την δημιουργία ενός ορισμού για τις τεχνητές μεθοδεύσεις και συμφωνούμε με τον εισηγητή. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα ε, για την ενημέρωση και σε πολλές σημεία θα χρειαστεί καλύτερη ε, πληροφόρηση όσον αφορά ε, την φοροαποφυγή και τις ε, εικονικές εταιρείες. Αντίθετα με το ΕΛΚ πιστεύουμε ότι ε, θα πρέπει να ενταθούν οι αρμοδιότητες και γι' αυτό θα πρέπει να προβληθεί και κάτι για την συμμετοχή και τη διαβούλευση των εργαζομένων. Αλλά αυτό θα χρειαστεί μια πιο λεπτομερή διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρτιν. Η Μπάρμπαρα Κάπελ δεν είναι παρούσα. Εκ μέρους του θέλετε το λόγο εσείς. Όχι. Θα δώσω πάλι το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Όλε Λούντιξον, για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για τις προτάσεις ε, που εξέφρασαν και για τις απόψεις που ε, εξέφρασαν. Θα συνεργαστούμε στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία με, τους απαραίτητους, με τις απαραίτητες συμβιβαστικές λύσεις. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι και να κινηθούμε προς την ίδια κατεύθυνση να βρούμε κάποια λύση σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Θα λάβω υπόψη μου λοιπόν ε, ε, τις απόψεις όλων των συναδέλφων και θα καταλήξουμε ελπίζω σε μια καλή λύση. Ευχαριστώ πολύ όλα. Προθεσμία για τροπολογίες είναι, 15η, ε, είναι η 5η Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα και θα συζητηθεί στις 8 και 9 Οκτωβρίου η έκθεση με τις τροπολογίες θα ψηφιστεί στις 18 Οκτωβρίου και θα ψηφιστεί στην Επιτροπή Γιούρη στις 19 Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι και τώρα εφόσον επανέρχεται ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη στις μισή, γιατί εκείνος θα προεδρεύσει στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης διακόπτουμε 5 λεπτά και θα αναλάβει ο κύριος Γκουαλτιάρης για αυτή την ε, σημαντική συζήτηση και να είναι παρόν από την αρχή της συζήτησης. Συνεχίζουμε λοιπόν στις 4 και 30.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 Καλώς λοιπόν συνεχίζουμε, πηγαίνουμε στο σημείο 19, έλεγχος ε, κατ' εξουσιοδότηση πράξεων και κατ' εφαρμογή αποφάσεων. Θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο SDS. Ο κανονισμός SDS, όπως ξέρετε, έχει τεθεί σε ισχύ τον μήνα Ιανουάριο από τις 17-18 Ιανουαρίου μέχρι αντίστοιχα τον Ιανουάριο του 19 και γι' αυτό είναι απαραίτητο να ληφθούν κάποιες αποφάσεις και κάποια μέτρα και ακριβώς θα συζητήσουμε ακριβώς τα θέματα των τεχνικών επιπέδων αναφοράς τα οποία έχουν προετοιμαστεί. Στην ουσία είναι μια μορφή ελέγχου, εν πάση περιπτώσει, της προπαρασκευής της Επιτροπής. Τα μέτρα αυτά αφορούν στην ΕΣΜΑ και την EBA, τεχνικά standards για την διαδικασία αδειοδότησης τρίτου μέρους σε σχέση με την συμμόρφωση, όπως επίσης και τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για την ομογένεια, ομοιογένεια ε, τους, των κινδύνων κατακράτησης. Υπάρχουν αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες. Νομίζω ότι η συζήτηση σήμερα είναι ενδιαφέρουσα. Καλωσορίζω τον Στίβεν Μάγιορ πρόεδρο της ΕΣΜΑ, τον Πίρς Χάμπεν, διευθυντή των τραπεζικών αγορών καινοτομίας και καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Πιστοτικής Αρχής και την Φελίσια Χανέσκου, Στανέσκου από πλευράς της Γενικής Διεύθυνσης φύσμα. E uh, Θα ακούσουμε λοιπόν την παρουσίαση για το RTS από πλευράς ε, της ε, Ευρωπαϊκής ε, Τραπεζικής Αρχής. Έχει ζητηθεί μια έγκαιρη υιοθέτηση και υποστηρίζω την πρόταση αυτή. Νομίζω ότι έχουμε προετοιμαστεί αρκετά για να σεβαστούμε αυτές τις προθεσμίες οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά πλέον. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρουσίαση του Μάιγιορ για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Ρομπέρτο που μου δώσατε το λόγο. Όπως ε, είπατε ήδη στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις, σε ένα τμήμα της προσπάθειας σε επίπεδο τεχνικό γενικά έχει ήδη ε, προχωρήσει. Ευχαριστώ την ΕΚΟΝ που μου δίνει την δυνατότητα να συμμετέχω σε αυτή την διαδικασία ελέγχου. Έχουμε ε, κάποιες βασικές ε, πλευρές ε, της δραστηριότητας της ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ όπως είπε ο Ρομπέρτο, ε, θα ξεκινήσουμε από την 1η Ιανουαρίου του 19 έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι των συνομοθετών ε, θα γίνονται σεβαστοί. Εγώ θα σας παρουσιάσω τις πρόσφατες δραστηριότητες της ΕΣΜΑ. Θα ξεκινήσω υπογραμμίζοντας τις βασικές αρχές που καθοδήγησαν τις ε, πολιτική της ΕΣΜΑ σε σχέση με την τιτλοποίηση και τη διασφάλιση ενός υψηλού επίπεδου διαφάνειας και προστασίας των επενδυτών στα πλαίσια των συναλλαγών τιτλοποίησης. Η ανάγκη για υψηλά επίπεδα διαφάνειας είναι το βασικό μάθημα που πήραμε από την χρηματοπιστωτική ε, κρίση. Πιστεύω ότι η αύξηση της διαφάνειας, της αγοράς τιτλοποίησης και οι διατομιακές συνεκτικές ρυθμίσεις και απαιτήσει θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη στην αγορά τιτλοποίησης και τις συναλλαγές γύρω από αυτή και θα βοηθήσουν τελικά ιδιαίτερα την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Τον Ιούλιο του 2016 η ΕΣΜΑ υπέβαλε το πρώτο σετ τεχνικών επιπέδων αναφοράς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κριτήρια λεγόμενα STS. και είναι υποχρεωμένοι λοιπόν όσοι συμμετέχουν στις συναλλαγές αυτές να ενημερώνουν την ΕΣΜΑ ότι οι συναλλαγές τους ανταποκρίνονται στα κριτήρια STS. Δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2018 και ένα δεύτερο σετ οδηγιών οι κανόνες αυτοί ε, δείχνουν ότι μια επιχείρηση όταν ζητά την αδειοδότηση για να αξιολογήσει τη συμμόρφωση μιας διαδικασίας ε, τιτλοποίησης πρέπει να χρησιμοποιεί και να βασίζεται στα κριτήρια STS. Ταυτόχρονα την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύσαμε και άλλη μία σειρά τεχνικών ρυθμίσεων για την ενημέρωση η οποία θα πρέπει να γίνεται στον τομέα των τυπλοποιήσεων. Όπως ξέρετε, ε, αυτά τα επίπεδα προστασίας θα εφαρμοστούν ήδη από τις 18 Ιανουαρίου του 2019. Όπως εξήγησα στην επιστολή που έστειλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συνομοθέτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει το πεδίο για να αποφύγουμε ε, μη απαραίτητες επιβαρύνσεις των συμμετεχόντων στις αγορές ε, μέσω της εφαρμογής των δύο σετ τεχνικών ρυθμίσεων. Οι πλατφόρμες αυτές είναι ιδιαίτερα λεπτομερείς, αλλά παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υιοθετήσει, να αντισυιοθετήσει το ταχύτερο δυνατόν η, Ευρωπαϊκή, η, αρχή ΕΣΜΑ κάνει προσπάθειες έτσι ώστε οι οδηγίες αυτές, τα μέτρα τα οποία προτείνει να βοηθούν στην σωστή διαφάνεια, την απαραίτητη διαφάνεια των συμμετεχόντων στις αγορές αυτές. Επίσης δίνουμε σε όλους τους ενδιαφερομένους τις απαραίτητες πληροφορίες και την δέουσα γενικά προφύλαξη και διαπιστώνουμε να, ότι υπάρχει ιδέουσα προφύλαξη στα πλαίσια των συναλλαγών τιτλοποιήσεων ιδιαίτερα σε διάφορους τομείς οι οποίοι μεταξύ τους δεν έχουν πάρα πολλά κοινά και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε με διαδροτικό τρόπο λόγω του υψηλού επίπεδου των λεπτομέρειας των, των οδηγιών αυτών είναι δύσκολο μερικές φορές να δούμε τι κριτήρια είναι αυτά τα οποία δεν μπορούν να γίνουν δημόσια. Αυτό δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα γιατί παλαιά δάνεια τα οποία πηγαίνουν καλά τώρα στατιστικά θα πηγαίνουν καλά και στο μέλλον αλλά αυτό σημαίνει ότι ε, οι προτινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν καταστάσεις όπου ορισμένα δεδομένα δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα βοηθήσει ε, να γίνουν κατανοητές σε συναλλαγές για τις οποίες δεν είναι επαρκή τα στοιχεία τα διαθέσιμα μέχρι τώρα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες δραστηριότητες στη ΣΕΣΜΑ παράλληλα με το λεγόμενο Single Roadbook, με το ενιαίο αυτό ε, οδικό χάρτη, έτσι ώστε να μπορούμε να δημοσιεύουμε τις σκηνοποιήσεις στον σωστό χρόνο στα πλαίσια ε, της ε, επίσημης σελίδας μας. Αυτή τη στιγμή εφαρμοστεί ε, η οδηγία τότε θα είμαστε σε μόνιμη επαφή με τους εθνικούς νομοθέτες και θα ελέγχουμε τις δραστηριότητες τους, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το ευρωπαϊκό πλαίσιο STS. Τέλος, στα πλαίσια των ε, εποπτικών μας ε, αρχών θα προσπαθήσουμε ε, να δούμε τι γίνεται και με τα καταθετήρια των ε, τιτλοποιήσεων. Ήδη από τον προϋπολογισμό του 19 όπως η δημοσιονομική διαδικασία για το 19 δεν έχει ολοκληρωθεί, ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει τις προτάσεις μας και τα αιτήματά μας έτσι ώστε να έχουμε τις δυνατότητες και τον χρόνο να ε, βοηθήσουμε σε ένα τόσο σημαντικό τομέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στίβεν. Και τώρα για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, EBA, ο Pierce happen. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, που μας καλέσατε για την ανταλλαγή απόψεων. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους της ΕΣΜΑ για την ε, αποτελεσματική εφαρμογή του ε, κανονισμού για την τιτλοποίηση. Η EBA έχει λάβει 29 εντολές ε, κανονιστικές ε, εντολές και φέτος εργαζόμαστε για έξι από αυτές ώστε να εξασφαλιστεί η ε, ομοιογενής εφαρμογή του, κανονισμού τυκλοποίησης. Τον, Ιούλιο ε, δημοσιεύσαμε δύο εντολές. Ο για την ομοιογένεια ε, ε, ε, ήταν αναμενόμενος στις αγορές γιατί αποτελεί το βασικό, τη βασική απέτυχη για την κρίση του STE αλλά και για την αξιολόγηση των υποκείμενων κινδύνων και γι' αυτό κατά τη σύνταξη του σχεδίου μελετήσαμε από τη, τη σκοπιά των επενδυτών για να δούμε εκείνοι πώς αξιολογούν το θέμα των κινδύνων. Τώρα, το σχέδιο RTS υπέστη εκταμένη συζήτηση και τη Κανονιστική επιτροπή και στον ιδιωτικό τομέα. Θα σα μεταφέρω τα βασικότερα θέματα. Για μας το πιο σημαντικό ήταν να υπάρξει επαρκή ισορροπία μεταξύ στου επαρκώ αυστηρού κανόνε που θα μα επιτρέψουν να προχωρήσουμε με την ομοιογενοποίηση ε, με βάση τι διαφορέ και τα χαρακτηριστικά των τυπλοποίησεων, αλλά από την άλλη πλευρά χρειάστηκε να δουλέψουμε για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είμαστε τόσο αυστηροί ώστε χωρί να το θέλουμε θέλουμε να ε, δημιουργήσουμε ε, συγκέντρωση, πράγμα που θα ευνοούσε τις τράπεζες με τους μεγάλους ε, ισολογισμούς. Και αν δείτε τον παράγοντα ομοιογενοποίηση θα δείτε ότι πετύχαμε την ισορροπία και κάναμε και προσαρμογή μετά τις διαβουλεύσεις για να το λάβουμε αυτό υπόψη μας. Πιστεύω ότι η ισορροπία πετέχθη τελικά. Επίσης θέλω να πιστήσω την προσοχή σας στους τέσσερις προϋποθέσεις της ομοιογενοποίησης που έχουμε ε, ε, ε, συγκεκριμενοποίηση στο RTS. Θέλουμε να εφαρμοστούν πλήρως για την εγγύηση και την ομοιογενοποίηση. Υπάρχει η απέτηση για τα χαρακτηριστικά της ταμιακής ροής και τέλος η απέτηση για την κατηγορία των, του ενεργητικού. Το άλλο σχέδιο αφορά την διακράτηση κινδύνου. Είναι κομμάτι της δουλειάς που έχουμε ήδη κάνει. Προσπαθούμε να μην ε, προκαλέσουμε ε, αναταραχή στην αγορά και θα ήθελα να σας πιστήσω την προσοχή σε διάφορες διατάξεις. Θα είναι πολύ πιο σαφές ότι όταν λέμε ότι ε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της πώληση ή του hedging, της ε, προστασίας, της μελλοντικής προστασίας και τελικά πιστεύω ότι κάναμε λειτουργική την απέτηση για την τιτλοποίηση των επιλεγμένων στοιχείων του ενεργητικού. Αυτό προσφέρει ε, νομική ασφάλεια και μια πιο εναρμονισμένη ε, εφαρμογή των κανόνων και άρα περιορίζει τη δυνατότητα του αρμπιτράς. Δουλεύουμε σκληρά για το επόμενο έτος ε, για το RTS του KIRB, τον υπολογισμό του KIRB και τον τον υπολογισμό της τίτλοποίησης από τους κεφαλαίου από τους επενδυτές. Κυρίως το πιο σημαντικό για μας φέτος και εκεί έχουμε επικεντρώσει την προσπάθειά μας είναι η δουλειά που έχει ξεκινήσει για τις κατευθυντές γραμμές της EBA για την ε, ε, ερμηνεία των κριτηρίων STS συνολικά. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα ενιαίο σημείο ερμηνείας αυτών των κριτηρίων και για τους χορηγούς και για τους επενδυτές αλλά και τις αρμόδιες αρχές και τους τρίτους, ε, τους πιστοποιητές. Συνεργαζόμαστε πολύ συχνά, ε, στενά με την ΕΣΜΑ και την ΕΑΙΟΠΑ για να εξασφαλίσει μια συνεπής και λειτουργική εφαρμογή των κανόνων που, ε, που προτείνουμε. Σας ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Η ενζωγόνηση της αγοράς της τυλοποίησης είναι σημαντική προτεραιότητα για μας, γιατί είναι σημαντικό στοιχείο ε, του θεματολογίου της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών. Το νέο πλαίσιο είναι ολοκληρωμένο και συνεπώς και πολύπλοκο. Το επίπεδο 1 έδωσε την εντολή στην Επιτροπή να υιοθετήσει κάποια ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και κάποια στοιχεία που αφορούν ε, και την αγορά τυπλοποίησης συνολικά. Καθαρά τεχνικά πρότυπα θα είναι σημαντικά ε, για το να γίνει λειτουργική η αγορά ε, τίτλοποίησης που είναι στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη και θα είναι σημαντικό και να διευκολύνουν ε, την ανάπτυξη όταν αρχίσουν ε, να είναι σε εφαρμογή οι κανόνες αυτή τον Ιανουάριο. Ιδιαίτερα για την τιτλοποίηση STS είναι σημαντικό να έχουμε τα τεχνικά πρότυπα για την ομοιογένεια. Αυτά τα οποία έχουν ετοιμαστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και τα πρότυπα τα οποία έχει προετοιμάσει η ΕΣΜΑ και όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι σημαντικό να έχουν ε, τεθεί σε εφαρμογή ε, οι κατευθυντήριες γραμμές ε, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών με τα κριτήρια που αναφέρθηκαν. Δύο σημεία είναι τα πιο σημαντικά. Τα τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις απαιτήσει για την αποκάλυψη πληροφοριών στους επενδυτές που έχουν ετοιμαστεί από την ΕΣΜΑ και ε, τα ε, κριτήρια ε, σχετικά με τον κίνδυνο και την απορρόφηση κινδύνου που έχουν διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Τώρα η Επιτροπή θα έχει το λόγο για πολλά από αυτά τα πρότυπα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρακολουθήσει το έργο των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Εργών και ευχαριστούμε τις εποπτικές αρχές για τη σκληρή δουλειά την οποία κατέβαλαν κατά τους περασμένους μήνες, συμπεριλαμβανομένων των καλοκαιρινών μηνών των διακοπών. Έχουν συνεισφέρει και εμπειρογνώμονες από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, έχουν γίνει πολλές διαβουλεύσεις ε, και ε, με αρμοδίους στο πλαίσιο ε, των αρμοδιοτήτων τους. Ε, έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες. Πολύ συχνά και πριν από τις προθεσμίες μας παραδόθηκαν τα κείμενα, ιδιαίτερα για την, τις απαιτήσει για την αποκάλυψη δεδομένων. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει 7 σχέδια τεχνικών, ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και προσπαθούμε να τα επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατόν. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Ε, κάποια μπορεί να μην είναι απαραίτητα για την λειτουργικότητα της αγοράς, αλλά η ταχύ εφαρμογή τους ε, και έγκρισή τους ε, θα είναι εξίσου σημαντική. Ευχαριστώ πολύ. Και πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, αναφέρεται και τον προϋπολογισμό και η ψηφοφορία που κάναμε σήμερα δεν ήταν πολύ θετική επ' αυτού. Θα προσπαθήσουμε όμως να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε την πρόταση της Επιτροπής. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Πολ Τάγκ. Πρώτη μέρα μετά τις διακοπές και μας υποδέχεται μία βροχή από κανονισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο το οποίο έχετε επιτελέσει στις ε, εποπτικές αρχές. Ε, ευχαριστούμε που ε, επιταχύνατε τις εργασίες σας, παρότι δεν έχετε πλήρη στελέχωση από ό,τι γνωρίζουμε. Είναι πολύ λεπτομερείς όλες αυτές οι διατάξεις και χρειάζεται η σωστή ισορροπία. Η γενική εικόνα που έχω είναι ότι ε, κινούμεθα προς τη σωστή κατεύθυνση ε, με σκοπό να αναπτύξουμε την αγορά της τυκλοποίησης. Έχω κάποιες ερωτήσεις, κυρίως βάσει των συζητήσεων που έχουμε κάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάποια σημαντικά θέματα. Δεν έχω εξετάσει όλες τις λεπτομέρειες, ε, αλλά πιστεύω βάσει των συζητήσεων που έχουμε κάνει ε, στο Κοινοβούλιο κάποια στοιχεία πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν ε, σαφείς απαιτήσει από τους τρίτους για τις ε, υπάρχουν κάποιες λειτουργικές εγγυήσεις που απαιτούνται, εγγυήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και η ερώτηση είναι πώς είστε βέβαιοι ότι αυτό το οποίο απαιτείται από ε, τρίτους όντως τηρείται στην πράξη. Αν αργότερα δηλαδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, Υπάρχει δυνατότητα να αποσύρεται η άδεια που δίδεται σε αυτούς τους τρίτους φορείς. Όταν κάναμε ε, τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, ανησυχούσαμε μήπως απλώς τους δίνετε την άδεια χωρίς να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές τους στη συνέχεια. Ένα άλλο σημείο τώρα για την αποκάλυψη στοιχείων. Πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχουν δεδομένα ή να μην είναι καλής ποιότητας τα δεδομένα. Πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα αυτό. Ιδιαίτερα όταν ο ισχυρισμός ότι δεν είναι διαθέσιμα τα δεδομένα είναι ένας τρόπος αποφυγής των προβλημάτων θα μπορούσαμε να βάλουμε ετικέτες, να βάλουμε πράσινο ε, ε, για τα, τις περιπτώσεις τις οποίες δεν χρειάζονται ε, υπερβολική έλεγχη για τα θέματα της τιτλοποίησης. Αν θέλουμε να δίνουμε πιο εύκολα διευκολύνσεις σε κάποιους που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουν υποβάλει ε, όλες τις πληροφορίες και ότι είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία, αν τους δίνουμε το πράσινο φως. Πώς είμαστε βέβαιοι ότι τα διαθέσιμα δεδομένα είναι πραγματικά διαθέσιμα και όντως καταλήγουν στις βάσεις δεδομένων των αποθετηρίων. Στο πρότυπο για την αποκάλυψη δεδομένων, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είναι κέριο για την ανάπτυξη της αγοράς, ε, κατά τι είναι διαφορετικό αυτό το πρότυπο από αυτά που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είμαι περίεργος για το πώς καταλήξατε αυτά, σε αυτά τα πρότυπα. Σχετικά με την ομοιογένεια, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που δεν έπρεπε να κάνουμε εμείς τη δουλειά, έπρεπε να την κάνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα χαρακτηριστικά του κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων. Και είναι δύσκολο να αποτιμήσουμε κατά πόσο τα κριτήρια ομοιογένειας για παρόμοια πρότυπα, για παρόμοιες διαδικασίες και υπηρεσίες, κατά πόσο συνεισφέρουν στα ίδια χαρακτηριστικά χρηματορροών. Θέλουμε δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μπαίνουν στο ίδιο πακέτο στοιχεία με διαφορετικό βαθμό κινδύνου. Να υπάρχει κάποια ομοιογένεια. Και όσον αφορά την απορρόφηση κινδύνου, ανέτρεξα στην αρχική νομοθεσία για να δω ποιο είναι το αρχικό κίνητρο. Είστε βέβαιοι ότι η απορρόφηση κινδύνου εδώ έχει το ίδιο κίνητρο όπως και στην αρχική νομοθεσία. Ε, και τα θέματα σχετικά με την αποκάλυψη νομίζω ότι είναι διαφορετικά ε, σε σχέση με την οριζόντια και κάθετη απορρόφηση κινδύνου. Μας ενδιαφέρει και η συχνότητα. Πόσο συχνά, με τι συχνότητα ετησίως έχετε τέτοιες περιπτώσεις ε, κάθε της απορρόφησης κινδύνου. Χρειάζεται κάποια ελάχιστη επεξήγηση των δεδομένων και θα θέλαμε να έχουμε και εμείς κάποια στοιχεία για την τιτλοποίηση. Ε, υπάρχει κάποιο αρμπιτράζ, πόσες ε, οριζόντιες, πόσες ε, κάθετες τέτοιες περιπτώσεις έχετε. Αυτό το οποίο θέλουμε όταν μιλάμε για την αποκάλυψη στοιχείων είναι να υπάρχει σωστή παρακολούθηση της αγοράς. ούτως ώστε να μην διατρέχει κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε τη σωστή παρακολούθηση, ούτως ώστε να μπορούμε παρακολουθώντας την αγορά να ξέρουμε ότι ε, επίκειται κάποιος κίνδυνος. Αυτά ήταν τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή για το ΕΛΚ εκ μέρους του κυρίου Κάρας στη, από τη διτή του ιδιότητα και σκιώδη και ως συγητή του CRR παρότι είμαστε για το συζητάμε το STS. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους που ήρθαν εδώ για την ανταλλαγή ιδεών και ζητώ συγγνώμη που ο κύριος Καράς ε, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί για ιατρικούς λόγους. Θα διαβάσω ε, λοιπόν τα σχόλια ε, και τις ερωτήσεις του. Καταρχήν, ως εισηγητής του, για τις τροπολογίες CRR για την ε, τιτλοποίηση και ως σκιώδης ε, του ΕΛΚ ε, για τον κανονισμό STS. Ο κύριος Καρά σας ευχαριστεί για την πολύ, για, για την πολύ κατάλληλη ευκαιρία που προσφέρετε σήμερα για τη συζήτηση. ο κύριος Καράς πιστεύει ότι στο επίπεδο 1 η διαφανής και ε, διασφαλισμένη, διασφαλισμένος έλεγχος είναι απολύτως απαραίτητος και θέλει να ρωτήσει αν υπάρχουν προβλήματα στο επίπεδο 1 που να επηρεάσουν το επίπεδο 2. Δεύτερον, ο κύριος Καράς ε, θεωρεί ότι είναι θετική η πρόοδος των πρόσφατων ε, προτάσεων για το RTS και το STS φυσικά πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω και γι' αυτό ζητά από, το, από τις, ε, τις ευρωπαϊκές αρχές της ESA να, ε, να μελετήσουν τις προτάσεις όσον αφορά το τελικό σχέδιο του RTS και ITS που πρόσφατα δημοσιεύτηκε. Ο κύριος Καράς έχει ε, τρεις ερωτήσεις προς τις ESA. Πρώτον για την ΕΣΜΑ, για το RTS και το ITS, για, την, για τις απαιτήσει αποκάλυψης. Όσον αφορά σχετικά με το σχέδιο ε, το, της αρχικής διαβούλευσης για το RTS, η, τα έντυπα αναφοράς δεν ε, θα εφαρμόζονται για την τιτλοποίηση. Όμως το τελικό σχέδιο του RTS μοιάζει ότι και αυτού του είδους η τιτλοποίη, όλες οι ιδιωτικές τιτλοποίησεις θα απαιτείται να αποκαλύπτουν τις ίδιες ε, ε, πληροφορίες όπως και οι δημόσιες τιτλοποίησεις. Είναι σωστή αυτή η αντίληψη και γιατί άλλαξε η ΕΣΜΑ το σχέδιο του RTS στο σημείο αυτό. Δεύτερον προς την EBA. Για το RTS για, την, για τα κριτήρια ομοιογένειας της, του STS. Υπάρχουν επιπλέον παράγοντες ομοιογένειας ε, που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις διαθέσιμες, τα διαθέσιμα πουλς για, την, για τις τιτλοποίησεις. Μήπως θα πρέπει ε, ένας παράγοντας ομοιογένειας να λαμβάνεται υπόψη και... E και μετά το EBA σχετικά με το RTS και για τη διακράτηση κινδύνου. Πρέπει να μας, θα θέλω να μας εξηγήσετε γιατί στο τελικό RTS το καθορισμένο spread των, δεν διατηρήθηκε στην επιλογή της διακράτησης. Τέλος, ο κύριος Καράς θέλει να ακούσει αν, να του πείτε εάν η Κομισιόν έχει ήδη απόψει σχετικά με την τροποποίηση των, το τελικού σχεδίου ρυθμιστικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΣΜΑ και η EBA. Οπότε, λέει ο Μιλήτρια, σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις που, οι οποίες θα διαβιβαστούν στον κύριο Κάρας και ζητώ συγγνώμη ε, που έπρεπε να τον ε, αντικαταστήσω. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρος. Uh, λοιπόν, δεν υπάρχουν μέλη από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Οπότε και εγώ μπορώ να θέσω κάποιες ερωτήσεις ιδιαίτερα στην uh, αρχή εποπτείας των τραπεζών Καταρχάς θέλω να συγχαρώ και την ΕΣΜΑ και την EBA για την δουλειά που έχουν κάνει μέχρι τώρα και σε σχέση με το RTS και το ITS. Είναι σαφές ότι υπάρχουν βέβαια πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να αναλύσουμε καλύτερα, αλλά νομίζω ότι οι προσπάθειές τους ήταν Μέχρι τώρα η πρώτη εντύπωση που έχω θετική. Ένα συγκεκριμένο σημείο για την ομοιογένεια δεν ξέρω αν υπάρχει μια σχετική, μια επιμέρους απόκληση ανάμεσα στην δήλωση αρχών και σε μια συγκεκριμένη παράγραφο του κανονισμού αρτίας, στο σημείο 42. Διευκρινίζεται είναι μια μακρά φράση, περίπλοκη, τα δάνεια μπορούν να θεωρηθούν προσφερόμενα προς τιτλοποίηση ακόμα και αν στην παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 3 του RTS υπάρχει μία αντίστοιχη δήλωση και δεν ξέρω εδώ τώρα αν η ανάγνωση η δική μου, η κατανόηση η δική μου είναι λανθασμένη. Αν υπάρχει μία διαφορά δηλαδή ανάμεσα στην παράγραφο 42 και στα συγκεκριμένα άρθρα. Πρέπει να υπάρχει απαραίτητη ομοιογένεια και ακόμα και όταν υπάρχει δεν υπάρχει μερικές φορές μηχανισμός ο οποίος να απο... υπάρχει μάλλον μια νομική ρύθμιση η οποία δεν επιτρέπει ουσιαστικά ομοιογενή δάνεια να συμπεριληφθούν ε, σε μια διαδικασία. Δεν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τώρα ποια είναι η άποψή σας γιατί όπως είπαμε στο άρθρο 20 Παράγραφος 8. Μιλάμε για ένα μόνο είδος, για ένα μόνο, για μία μορφή ενεργών. Δεν ξέρω λοιπόν αν υπάρχει μία διαφοροποίηση, θα ήθελα την άποψή σας γύρω από αυτά. Περβάνς θες κάτι να προσθέσεις. Ο Στίβεν είναι ο πρώτος που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ για τις σκέψεις τις οποίες εξέφασαν τα μέλη σας. Είναι κατανοητό ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αξιολογήσετε τη δουλειά την οποία έχουμε κάνει, αλλά οι αρχικές σας παρατηρήσεις ήταν θετικές κάποια σχόλια πάνω στα σημεία τα οποία έθεσαν τα διάφορα μέλη της Επιτροπής σας. Πρώτον, ε, για τους πίνακες ε, οι οποίοι... And I should say here, obviously we have uh, built our work. Είναι προφανές ότι έχουμε εμείς βασιστεί στους υπάρχοντες πίνακες και στην δουλειά που έχει ήδη υπάρξει. Ξέρουμε τους αντίστοιχους πίνακες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας. Είναι η βάση την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει ε, για τα τεχνικά μέτρα τα οποία έχουμε ήδη δημοσιοποιήσει. Υπάρχουν ταυτόχρονα νέες απαιτήσεις στον κανονισμό που θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται εδώ. Ο νέος κανονισμός είναι πιο σαφής για την προστασία των δυνητικών επενδυτών όπως επίσης και των δημοσίων αρχών να είναι σε θέση να δείχνουν να είναι βέβαιοι για την, πριν πάρουν κάποιες αποφάσεις την απαιτούμενη προσοχή και βασικά χρησιμοποιούμε ακριβώς ένα είδος μέτρων τα οποία χρησιμοποιούσαμε και στο παρελθόν Ταυτόχρονα όμως έχουν υπάρξει κάποιες προσθήκες, έχουν υπάρξει κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις. Υπήρξαν ερωτήσεις επίσης και για τη σχέση ανάμεσα στις δημόσιες τιτλοποιήσεις και τις ιδιωτικές τιτλοποιήσεις. Επ' αυτού, εμείς και σε πρώτο επίπεδο και στα πλαίσια της προσεκτικής ανάγνωσης που κάναμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχει παρά πάρα πολύ μικρή δυνατότητα να γίνει η διάκριση ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα γύρω από τα θέματα τιτλοποίησης και την υποχρέωση δημοσιοποίησης. Είναι προφανές ότι θα υπάρξουν διαφορές σε σχέση με τη δημόσια ενημέρωση, αλλά η ενημέρωση που θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται με τους επενδυτές, με συγκεκριμένους επενδυτές, δεν διαφοροποιείται στο επίπεδο 1. Θα προτιμούσα να υπήρχε μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση, αλλά πάντως εμείς το κάνουμε αυτό λόγω ακριβώς ε, του επίπεδου α, του πρώτου επίπεδου. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι υπάρχουν λιγότερες δεσμευτικές υποχρεώσεις εδώ για τον ιδιωτικό τομέα. Μια άλλη ερώτηση αφορά τις αδειοδοτήσεις των τρίτων νερών που ε, προσφέρουν εγγυήσει σχετικά με τα κριτήρια του STS. Αυτό το οποίο κάνουμε εμεί σε τεχνικό επίπεδο, σε επίπεδο τεχνικών μέτρων, είναι γύρω από τις ενημερώσεις οι οποίες θα πρέπει να δίδονται προς τον εθνικό νομοθέτη ε, και να υπάρχει όπως είπα σε μια πρώτη φάση εποπτεία σε εθνικό επίπεδο και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πλαίσια βέβαια της διαδικασίας και της λογικής σύγκλησης που μας χαρακτηρίζει και εμείς κάνουμε εδώ αξιολογήσεις υψηλού επίπεδου. Είναι και αυτή μια δύσκολη προσπάθεια. Ταυτόχρονα έχουν υπάρξει αρκετές διαβουλεύσεις και έχουμε ασχοληθεί ε, με συγκεκριμένα παραδείγματα για να δούμε ακριβώς τι είδους ε, πληροφορίες και στοιχεία λαμβάνουμε υπόψη όπως ακριβώς ε, και για τις υπηρεσίες αξιολόγησης. Έχουμε εμπνευστεί από την εμπειρία που έχουμε σε άλλους τομείς οπότε στα πλαίσια της, των συγκλίνουσών εποπτικών δραστηριοτήτων μας προσπαθούμε να προχωρούμε σε ουσιαστικές αξιολογήσεις για τα θέματα της ποιότητας των δεδομένων και σε ποιο βαθμό είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε κάποια πράγματα όταν δεν είναι διαθέσιμα τα δεδομένα και τι σημασία έχει η δημοσιοποίηση στοιχείων προς τα έξω. Ξέρουμε εμείς πόσο προβληματική ήταν ε, στην περίπτωση της χρηματοπιστωτικής χρήσης η έλλειψη ενημέρωσης και στα πλαίσια των τιτλοποιήσεων. Γνωρίζουμε όμως και αναγνωρίζουμε ότι ορισμένα στοιχεία δεν μπορεί να δημιουργούνται Παλαιά δάνεια σαν παράδειγμα για τα οποία δεν είχαμε τις πληροφορίες αυτές. Αν υπήρχαν ε, θα μπορούσαν φυσικά να ζητηθούν σαν στοιχεία αξιολόγησης πιθανής τιτλοποίησης. Κάναμε λοιπόν μία αξιολόγηση για να προσπαθήσουμε να δούμε εάν είναι θεμητό τέτοιου είδους πληροφορίες να θεωρούνται ως μη διαθέσιμες και αν πράγματι υπάρχει η δυνατότητα να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους υπάρχει αυτή η μη διαθεσιμότητα των στοιχείων. Γι' αυτό ακριβώς στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης πλατφόρμας λέμε ότι δεν είναι δυνατόν να κανείς να αποκλίνει και έχοντας περισσότερες εμπειρίες μπορούμε να αυξήσουμε το επίπεδο των προσδοκιών για το τι είναι διαθέσιμο και τι όχι. Και το προτελευταίο σχόλιο μου και υπήρξε μια ερώτηση αν όλα πάνε καλά. Ναι, προς το παρόν εμείς πιστεύουμε ότι και τα υπόλοιπα τα οποία θα ανακοινώσουμε θα έρθουν έγκαιρα. Περιμένουμε και από την EBA τις διαδικασίες για το clearing. Εδώ υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση. Έπρεπε ε, εμείς να τα δημοσιεύσουμε αυτά πριν το καλοκαίρι ε, στα πλαίσια του τρίτου τετραμήνου. Αλλά Ελπίζω ότι όλα τα άλλα πηγαίνουν έγκαιρα. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω αυτό που λέμε για τον προϋπολογισμό. Αν δεν έχουμε τον προϋπολογισμό που θα μας επιτρέψει να εποπτεύουμε, δεν θα εποπτεύουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό από μακράν. Είναι σαφές ότι έχουμε ανάγκη από συγκεκριμένους ανθρώπινους πόρους Μπορούμε ίσως μία χρονιά να καλύψουμε κάποιες ελλείψεις που έχουμε στα πλαίσια της μηδενικής αύξησης των ανθρώπινων πόρων που είναι στη διάθεσή μας, αλλά υπάρχουν υπηρεσίες που ελέγχουν τον προϋπολογισμό μας και ελέγχουν και αυτές ότι έχουμε ανάγκη ακριβώς από μια καλύτερη, ε, μεγαλύτερη άνεση. Τώρα, θα υπάρξουν λοιπόν για τις τιτλοποιήσεις πολύ περισσότερες ενημερώσεις και πληροφορίες έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτά τα οποία συνέβησαν με τις τιτλοποιήσεις κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Είναι μία επιπλέον αλλαγή αυτή σε σχέση με το παρελθόν. Να υπενθυμίσω ότι ο κανονισμός για την τιτλοποίηση απαιτεί να υπάρξει ε, μια σωστή παρακολούθηση της αγοράς τιτλοποίησης στον σωστό χρόνο, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τους συνομοθέτες, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ, πολύ. πολύ. Ε, υποβλήθηκαν κάποια πολύ καλά ερωτήματα. Θα στραφώ σε αυτά ε, καταρχήν το θέμα του, ε, των χαρακτηριστικών ε, του, της ταμιακής ροής. Αυτή είναι ακριβώ η ισορροπία που είχα αναφέρει. όσον αφορά την ταμιακή ροή, η, ε, η συνέπεια της, της εξυπηρέτησης καλύπτει αυτό και εν πάση περιπτώσει φροντίζουμε να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα. Το απόλυμα είναι μπορεί κανείς να διακρίνει μετα μεταξύ του prime και του subprime σαφώ όχι. Μπορεί κανείς να είναι... Μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Να, να φτάσει σε περισσότερε λεπτομέρειες βεβαίω. Αλλά τελικά σε αυτό καταλήξαμε. Αν το ερώτημα είναι ε, μεγαλύτερη, αφορά τη μεγαλύτερη εικόνα, ναι. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της, το θέμα της συνθετικής διακράτησης, ε, ενδιαφέρον, θα το συζητήσουμε στο CORB, στο CURB και αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα, υποβα... θα δημοσιεύσουμε νέες απαιτήσει για τις αναφορές της τιτλοποίησης την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να καταλάβουμε το είδος της διακράτησης που υπάρχει, αν μπορεί να βελτιωθεί ή όχι, είναι αρκετά ενδιαφέρον, το συζητάμε και μελετάμε τα δεδομένα. Επίσης, ερωτήσεις για την ομοιογένεια, αν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τουλάχιστον ότι ένας τουλάχιστον τέτοιος παράγων πρέπει να λαφθάνει την υπόψη. Ναι, αν έχουμε τώρα ε, όρια ε, συνάφειας, materiality, ναι, υπάρχουν. Και όσον αφορά το spread, για μας το θέμα ήταν ότι αυτό δεν συμπεριλαμβανόταν στο προηγούμενο πρότυπο. Είπα ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε συνέχεια στο, σε αυτό που κάνουμε όσον αφορά τη διακράτηση κινδύνου. Και το τελευταίο ερώτημα του Προέδρου που είναι το πιο δύσκολο <laughs> και σύνθετο. Η ουσία είναι ότι έχουμε φτάσει στο άρθρο 20 να έχουμε ένα παράγοντα ομοιογένειας. Μπορεί κανείς να έχει είτε χαμηλό, ή χαμηλή κατάταξη ψηλη άρα δεν γίνεται ανάμειξη και άρα νομίζω ότι το καταφέραμε αυτό. Thank you. Um, so you, so Ευχαριστώ. Λέτε ότι η διατύπωσή σας συμβαδίζει με το άρθρο 42. Μάλιστα. Νόμιζα ότι δεν ήταν, αλλά αφού το λέτε. Θα το δω και μπορεί να επανέλθουμε. Ο εισηγητή. Α, όχι, όχι, συγγνώμη, ξέχασα να δώσω λόγο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Δεν θα σας καθυστερήσω. Αναφερθήκαμε όμως ως Επιτροπή σε δύο παρατηρήσεις. Στα σχολεία του κυρίου Κάρας Μα ζητήθηκε να πούμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση. Και η απάντησή μας είναι ότι προσπαθούμε να προχωρήσουμε το δυνατόν ε, ταχύτερα με βάση τα όσα έχουμε λάβει για τα πρότυπα. Συνεργαζόμαστε σε τεχνικό επίπεδο πολύ στενά με τις ε, ε, εποπτικές αρχές. Συμφωνούμε με τη γενική τάση των σχεδίων, αλλά χρειάζεται να γίνει νομική εξέταση των σχεδίων και αυτό χρειάζεται χρόνο. Και θέλω να απαντήσω και σε ένα άλλο σημείο σχετικά με την αποκάλυψη στοιχείων για τις ε, ιδιωτικές συναλλαγές. Ξέρω ότι έχει συζητηθεί το θέμα. Καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό. Δηλαδή, ότι η αποκάλυψη στις εθνικές αρμόδιες αρχές θα είναι το ίδιο και για δημόσιες και για ιδιωτικές συναλλαγές, αλλά η αποκάλυψη προς το κοινό είναι πιο περιορισμένη για τις ιδιωτικές συναλλαγές και νομίζω ότι αυτή η συμβαστική λύση είναι σχετικά ε, σωστή και δικαιή. Ευχαριστώ πολύ. Άλλα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας που ήρθαν στην Επιτροπή μας και που επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να ε, συνεργαστούν μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να ε, είμαστε ευθυγραμμισμένοι και με την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Η καταψήφιση της τροπολογίας επανέφερε το κείμενο του Συμβουλίου. Ήταν αντίθετο με τη λογική της πλειοψηφία που απέριψε αυτή την τροπολογία. Είναι ένα τεχνικό σημείο που νομίζουμε ότι θα το επαναφέρουμε. Με τη διατύπωση θα προσπαθήσουμε στο διάλογο που θα ακολουθήσει με τους φίλους μας της Επιτροπής Προϋπολογισμών να επαναφέρουμε το σημείο αυτό για να είμαστε συνεπείς ε, όσον αφορά τα καθήκοντα που σας αναθέτουμε και τους πόρους που πρέπει να έχετε για να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την παρουσίαση και για τις εξηγήσεις που μας δώσατε και θα συνεχίσουμε το διάλογο μέχρι την τελική έγκριση των προτύπων από την Επιτροπή. Νομίζω τώρα ότι ολοκληρώσαμε τη συνεδρίασή μας. Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα είναι η επόμενη συνεδρίασή μας. Πέρα στη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ.